πλαίσια των ευρωεκλογών είναι θέμα που θα ζητήσει σήμερα στις 5 και 10, στο 17 η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης της ε, εκ νέου χρήσεως των πληροφοριών δημοσίου τομέα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις να εγκρίνουμε το σχέδιο έχουμε όλες τις γλώσσες για διερμηνία. Εκτός από κρατικά δανέζικα, μαλτέζικα, λετωνικά και κελτικά. Τώρα έχουμε τις κατανάθεση πράξεις, τις εφαρμοστικές πράξεις και θα σας διαβάσω την σειρά αυτών εφαρμοστικές. Η Γραμματεία έχει διανύμει την εφαρμοστική απόφαση ε, για τον κανονισμό του 2016 του Κοινοβουλίου και αφορά την επαρκή προστασία προσπαθωμένων από την Ιαπωνία. Αυτό είναι η εργασία το οποίο έχει τις σχετικές ε, τροποποιήσεις του κειμένου. Ε, αυτά θα συζητηθούν ατύπως, τα έχουν συντάξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα λάβετε τα έγγραφα στο δελτίο τύπου μας, 16-18, η δε ε, ε, προθεσμία για ενστάσεις εδώ στην Λίμπε ήταν 23-18 το μεσημέρι και ε, αν δεν έχετε λοιπόν κάποια ένσταση να το υποβάλλετε μέχρι την προθεσμία και θα γίνει ψηφοφορία με τις ηλεκτρονικές κάρτες αύριο στις 9 και 4 να πάρετε την κάρτα σας και τώρα κάποιοι από τους συναδέλφους είναι στο δρόμο προς τα εδώ. καιρό Δευτέρα, βλέπετε. Ο κόσμος πολλές φορές αργεί να φτάσει με τα μέσα συγκοινωνίας. Αλλά μπράβο σε αυτούς που τα κατάφεραν να έρθουν καιρός. Στο τρία τώρα, συνάδελφοι. Να σας πω τα της παρακολούθησης της διαδρομής της ακρόασης για την νεολαία στην Ευρώπη. Ευτυχώς το μεταδίδεται από το ε, δίκτυό μας στο ίντερνετ στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για την εκδήλωση αυτή. Καλώς όρισαν επομένως οι νέοι και νεαροί ομιλητές μας από την ε, Σχολή Επιχειρηματικών Σπουδών Φόρεν ή Τόρεν. Και επίσης ε, να χαιρετήσουμε και αυτούς που μας παρακολουθούν από το ίντερνετ, από τα μέσα δικτύωσης και όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει στην συζήτηση στο hashtag 2018. Θα το δείτε και στην ε, οθόνη, αν δεν το είδατε ήδη, στην οθόνη που έχουμε στην αίθουσα. Αυτά όσον αφορά τη σχετική διαδικτυακή συζήτηση. Και όπως τα γνωρίζετε, αυτή η εκδήλωση που το ονομάζουμε I, για συντομία, έγινε πρώτη και δευτερήνη του 18, συμμετέσχουν 9.000 νέοι Ευρωπαίοι που συζήτησαν σε τέτοιους για μια καλύτερη Ευρώπη. Αυτό έγινε στο κοινό στο Στασβούργο. Πάρα πολύ εντυπωσιακή ήταν η εκδήλωση και σήμερα ε, κάνουμε αυτήν την ε, ε, συνέχιση της εκδήλωσης εκείνης, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα σχετικά με εκείνη την ε, εντυπωσιακή εκδήλωση θα έχουν κάποια απτή συνέχεια και ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου πρόκειται να λάβουν υπόψη τους όσα έχουν συζητηθεί και θα συζητηθούν. Άρα, σήμερα είναι η δεύτερη από 7 που έχουν προγραμματιστεί στη συνέχεια του 2018. Οπότε, σήμερα θα ακούσουμε ιδέε που έχουν σχέση με τα θέματά μας, αλλά θα πρέπει και να τοποθετηθούμε σε σχέση με όσα ακούσουμε και έτσι να κάνουμε κάτι που να αποτελεί πολιτική ε, τοποθέτηση και αντίδραση. Έχουμε εδώ δραστήριους έμπειρους συναδέλφους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση και άλλοι που θα έρθουν ε, σύν το χρόνο. Τώρα, οι τρεις νέοι πρόκειται σήμερα να μας προσέχουν τις ιδέες τους και αποδέκτες των προτάσεων αυτών θα είναι οι ευρωβουλευτές. Άρα, περί ιδιών, ο λόγος σήμερα. Όπως λέει το κείμενό μας, ο καθένας από τους νέους μας πρόκειται σε δύο λεπτά να κάνει την παρεμβασή του και οι συνάδελφοι, εάν δεν είναι πολύ κουρασμένοι από το ταξίδι τους για να έρθουν εδώ, θα πρέπει να τοποθετηθούν αν έχετε την απαραίτητη ενέργεια, να τοποθετηθείτε, να αντιδράσετε. Δύο λεπτά. Και εσείς δύο λεπτά, όποτε τώρα. Τι ζητήματα θα θίξουμε πολύ σημαντικά θέματα της Επιτροπής μας. Πρώτα-πρώτα η μετανάστευση. Και θα εστιαστούμε πιο συγκεκριμένα στους ασυνόδευτους ανηλίκους, στον ρόλο των μεταναστών, στην ε, κοινωνία των πολιτών, στην ε, πολιτική ένταξη και κατά δεύτερο λόγο θα δούμε προτάσεις για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Ωραία, ας ξεκινήσουμε τώρα με τους ε, τρεις νέους από το ΆΕ 2018. Λούκας Φόκτερ, Ραχίλ Τζανφάνια και Σιμών Έμπερς. Καλώς ορίσατε στην ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Αρχίζουμε με το πρώτο θέμα, τη μετανάστευση και όπως είπαμε να σταθούμε στους εσνοδούς ανηλίκους, στο ρόλο των μεταναστών στην κοινωνία και Από ό,τι γνωρίζω πρώτη θα μιλήσει η Ρέιτσελ. Με τις δύο προτάσεις της όσον αφορά την ε, παιδεία ε, και την επιμέλεια των πλαισίωση των ε, ανηλίκων, των εσνοδεύτων και που έχουμε γενία. οικογένειε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Μεταξύ τη 1 η Ιανουαρίου και τη 31 η Μαρτίου 2018, 927 συνόδευτα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά του φτάσαν στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης. Τα παιδιά αυτά δεν ζητούν ελεημοσύνη, αλλά θέλουν ευκαιρίε και πραγματικέ δυνατότητε για να συμμετάσχουν στην κοινωνία των πολιτών. Η πρώτη μου λοιπόν ιδέα ήταν να δώσουμε στα παιδιά αυτά, αλλά και στου νέου μετανάστε και πρόσφυγε, ευρωπαϊκέ υποτροφίε προκειμένου να μπορούν να πάνε άμεσα στο σχολείο, καθώ επίση και μια ισότιμη αναγνώριση των διπλωμάτων διπλωμάτων ή ένα σύστημα συγκριτική αξιολόγηση των διπλωμάτων και αυτό να γίνεται με τον πιο γρήγορο, φτηνό και εύκολο τρόπο. Θα πρέπει να, να δημιουργηθεί ένα νέο ταμείο προκειμένου όλα αυτά τα παιδιά να μπορούν να ενταχθούν στα ευρωπαϊκά σχολεία. Αυτό θα πρέπει να γίνει επίση και για του νέου μετανάστε προκειμένου να συνεχίσουν ή να αρχίσουν τι σπουδέ του. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να συνοδεύεται από πιο γρήγορε διαδικασίε που θα παρέχουν προστασία από τι εθνικέ αρχέ προκειμένου να μπορούν οι νέοι αυτοί και τα συνόδευτα παιδιά να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση αναμονής περιμένοντας να νομοποιηθεί η παραμονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα αυτόματο σύστημα ισοδυναμίας διπλωμάτων ή συγκρατικής αξιολόγηση των ήδη αποκτηθέντων διπλωμάτων και κατά αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί επίσης και το δίκτυο για τα Εθνικά Κέντρα Πληροφοριών για την αγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων και θα μπορούν όλοι αυτοί οι νέοι τα παιδιά να αντεχθούν σε σχολεία και πανεπιστήμια. Το πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκό, θα πρέπει να ασχολούνται με αυτό όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει όλες οι χώρες να συμβάλλουν προκειμένου παιδιά και συνόδευτοι ενήλικοι να μπορούν πραγματικά να ενταχθούν σε σχολεία πανεπιστήμια προκειμένου να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να τα βοηθήσουμε να εξελιχθούν στο μέλλον και να καταπολεμηθεί οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση. Πρόκειται για μια αμοιβαία υποφελή διαδικασία. Όπω είπε η Μισελ Ομπάμα, τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν σχολείο συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ ανεξάρτητα από το καθεστώ του, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του. Το να ανοίξουμε τι πόρτε των σχολείων και των πανεπιστημίων μα στα ασυνόδευτα, συνοδευόμενα και τα παιδιά τα οποία έχουν αποχωριστεί τι ε, οικογένειέ του, καθώ επίση και στου νέου μετανάστε, ουσιαστικά θα βοηθήσει να αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μα ιδρυμάτων και στην ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας. Η πρακτική αυτή θα δημιουργήσει μια ενάρετη θετική συνεργασία μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων, μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών και θα δώσει κατά αυτόν τον τρόπο σε όσους φεύγουν από τη χώρα τους και δεν μπορούν να ακολουθήσουν νόμιμες οδούς μετανάστευσης τη δυνατότητα να συνεχίσουν τουλάχιστον τις σπουδέ τους. Η δεύτερη μου ιδέα έχει να κάνει με το δικαίωμα των παιδιών στην αψυχή, το παιχνίδι και τη μελέτη. Είμαι εκπαιδευόμενη δικηγόρος από από την Ιταλία. Εξειδικεύομαι στο ζήτημα του ανθρωπίνου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κοινωνικού δικαίου και θεωρώ ότι θα πρέπει το δικαίωμα αυτό στην αψυχή και τη μελέτη να ισχύει για όλα τα παιδιά και για τους νέους μετανάστες και τα συνόδευτα παιδιά μετανάστες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ασχοληθούμε λοιπόν με το ζήτημα της επιμέλειας των μη συνοδευόμενων αυτών παιδιών προκειμένου να καταφέρουν να ταχθούν σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρμονίσει την εθνική νομοθεσία όσον αφορά τα εκτοπισμένα παιδιά, προωθώντας την βέλτιστη πρακτική του να μπορούν τα παιδιά αυτά να εξακολουθούν να ζουν σε ένα οικείο περιβάλλον από την εντάσσονται αυτόματα σε κέντρα για ανήλικους, όπου εκεί δεν τηρείται πάντα ω απόλυτη προτεραιότητα το μείζον συμφέρον του παιδιού. Απόλυτο στόχο τη επιμέλεια πρέπει να είναι η βαθύτερη ένταξη των παιδιών στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αναφερόμαστε μόνο στα συνόδευτα παιδιά όταν μιλάμε για επιμέλεια, αλλά και για του εκτοπισμένου γονεί, του γονεί μετανάστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε κοινού κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν έχουμε ένα σύστημα επιμέλεια για τα συνόδευτα παιδιά αλλά και για του εκτοπισμένου γονεί, δημιουργείται μια αμοιβαία εποφελή ε, νομοθεσία. Μπορούν τα παιδιά να ενταχθούν σε μια οικογένεια που θα τα φροντίσει και από την άλλη εκτοπισμένοι γονεί του, οι μετανάστε γονεί του, να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να βρουν ένα σπίτι, να καταφέρουν να ενσωματωθούν περισσότερο στην οικογένεια. Τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε μελέτη αλλά και σε αναψυχή και κατά αυτόν τον τρόπο πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ οικογένειε θα μπορέσουν να ασχοληθούν, να παράσχουν επιμέλεια στα παιδιά των μεταναστών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα επιμέλεια τέκνων λαμβάνοντα υπόψη ότι οι επενδύσει των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδώσουν πολύ περισσότερο από το να τοποθετηθούν πολύ απλώ τα παιδιά σε κάποια κέντρα για ανήλικου. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σύστημα πολύ πιο άμεσο, χωρί διαμεσολαβητέ και χωρί όλε τι ενδιάμεσε δαπάνε που συνήθω προκύπτουν. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα συνοδευόμενα, μη συνοδευόμενα παιδιά και τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τι οικογένειέ του θα καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τι δυνατότητέ του, θα μπορέσουν να μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι πραγματικές τους ανάγκες θα την χάνουν πλήρου ικανοποίηση και όπου αυτό το οποίο θα προέχει πάντα θα είναι το μείζον συμφέρον του παιδιού. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρέιτσελ. Δεν είναι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. Μπορείτε να χειροκροτήσετε βέβαια αν θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, δυνατότητα που μας δώσετε να παρακολουθήσουμε τις δύο αυτές ιδέες σας. Προτού τη δράσουν οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές θα ακούσουμε και τον Λούκας ο οποίος ε, θα μας μιλήσει για τη δυνατότητα διαμονής των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αξιόπιστοι ευρωβουλευτές ε, που μας καλέσατε. Η πρώτη ιδέα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η Ευρωπαϊκή Διαπαραμονή για άτομα με υψηλά προσόντα. Μιλάμε βεβαίω για την οδηγία της μπλε κάρτας η οποία υπάρχει ήδη αλλά δεν έχει καμία πρακτική χρήση. Η Κομισιόν ήδη προσπάθησε να τη μεταρρυθμίσει το 2016 αλλά απορρίφθηκε αυτή η προσπάθεια με βασικό επιχείρημα ότι η μετανάστες θα πρέπει να είναι στα χέρια των κρατών μελών. Κάτι με το οποίο συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι μια ομάδα πλήττεται ιδιαίτερος από την οδηγία της μπλε κάρτας. Οι νέοι από ολόκληρο τον κόσμο που ήρθαν και σπούδασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το άρθρο 5.3 της σχετικής οδηγίας λέει ότι για μια μπλε κάρτα χρειάζεται μία μισή φορές ο μέσος ετήσιο ετήσιος μισός της χώρας. Ε, εγώ είμαι από την Αυστρία, δηλαδή ο μέσος ε, καθάριστος μισθός ε, του 2016 ήταν 31.000 ευρώ. Θα τελειώσω την νομική του χρόνου και αμφιβάλλω αν θα μπορέσω να βγάζω 46.000 ευρώ όταν ξεκινήσω να δουλεύω. Οπότε προτείνω να προσθεθεί μια εξαίρεση στο άρθρο 5.3 για άτομα τα οποία αποφυτούν, φίτησαν και αποφυτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν έχει νόημα οικονομικά να εκπαιδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους και όταν είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία να βοηθήσουν να δημιουργήσουν τους διώχνουμε. Να δοθεί δηλαδή μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους ε, να λάβουν και αυτή μέρος ε, στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Διόδες. Μια μικρή αλλά αποτελεσματική αλλαγή. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε για την νόμιμη μετανάστευση. Ήδη δύο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. σε θέματα που αφορούν το νομοθετικό μας έργο. Είναι λίγο άδικο βεβαίω γιατί ξέρω πως ήρθαν λίγο αργά οι βουλευτές που ενδιαφέρονται. Βλέπω λοιπόν την Άννα Μαρία και την Σεσίλ να δω αν μπορούν να απαντήσουν. Λοιπόν, θα ζητήσω από την Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ πρώτα να απαντήσει, μετά από την κυρία Κιέγγι και μετά από τον Μπόντο Βαλέρο. Ευχαριστώ Κλοντ. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, καθυστέρησε το αεροπλάνο μου και να καλωσορίσω και τους νεαρούς εκεί στο βάθος. Ε, πραγματικά χαρά μας ε, το ότι επιτρέπεται σήμερα η Επιτροπή μας να γίνει το σπίτι των νέων της Ευρώπης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ιδιαίτερος που είχα ευκαιρία να σας ακούσω. Να σας πω ότι με την συνάδελφο την Κατερίνα Κινίτσι Ιδρύσαμε την διακομματική αυτή ομάδα των παιδιών, των, ε, για τα δικαιώματα των παιδιών, των νεαρών, έτσι ώστε να ενταχθεί σε όλο το νομοθετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ιδέα ότι το παιδί είναι πρώτα απ' όλα παιδί ανεξαρτήτως ε, του νομικού καθεστώτος κτλ. Και νομίζω ότι καταφέραμε χάρη στους συναδέλφους μου να έχουμε μια ισχυρή πλειοψηφία που να ξεπερνά τις πολιτικές ομάδες ε, με σκοπό τα συμφέροντα του παιδιού, ειδικά στο πακέτο ασύλου και μετανάστευσης. Ε, δυστυχώς όμως έχει παγώσει στο Συμβούλιο αυτή η μεταρρύθμιση όλες, όμως οι τροπολογίες ε, πέρασαν και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τους ε, συναδέλφους για αυτά τα οποία είπατε πράγματι ένα παιδί, όλα τα παιδιά, τα συνόδευτα μετανάστες ετούντες άσυλο πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε εκπαίδευση και σχολεία. Η Ευρώπη θα πρέπει να σημαίνει ασφάλεια για όλα τα παιδιά και πρόσβαση στα σχολεία και την εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ένταξη και να διδάξουμε και τις αξίες μας και να τους δώσουμε την ευκαιρία να οικοδομήσουν ένα νέο μέλλον στην Ευρώπη. Το άλλο θέμα, το θέμα των ανάδοχων οικογενειών, ναι, και αυτό είναι κομμάτι του πακέτου ασύλου, το δικαίωμα στο παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, έχουμε ζητήσει στα κέντρα υποδοχής να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ένα σημείο που μπορούν να παίξουν τα παιδιά με ασφάλεια. Επίσης έχουμε περιλάβει ε, κάποιες ε, διατάξεις για τη φυσική κυριότητα των κοριτσιών από τους ε, παιδικούς ε, γάμους, την τον γενετικό ακροτηριασμό, που τα οποία βέβαια πέρα από εγκλήματα εμποδίζουν και τις ίσες ευκαιρίες. Ε, να αναφέρω κάτι στον Λούκας που ανέφερε την παραθμισή της μπλε κάρτας μαζί με την συνάδελφο την... και ε, κοιλία. Περάσαμε νομοθεσία για την πρόσβαση των υπηκών τρίτων χωρών για στόχους κατάρτισης, εκπαίδευσης, έρευνας. Είναι λοιπόν μια επιταχυμένη διαδικασία για να σπουδάσουμε στην Ευρώπη και να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα ταλέντα γιατί συχνά σπουδάζουν στην Ευρώπη και πηγαίνουν στην Αμερική. Οπότε για να κρατήσουμε αυτά τα ταλέντα γιατί είμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να κερδίσουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τα ταλέντα στην Ευρώπη. Το τέλος καταφέραμε να υπερψηφίσουμε ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να κρατούνται ε, λόγω του νομικού καθεστώτος τους όταν έρχονται στην Ευρώπη. Ε, πρέπει να έχουν αντιμετώπιση όπως ε, και τα παιδιά με ευρωπαϊκή υπηκότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Άννα Μαρία. Θα πρέπει να τηρούμε όμως το χρόνο αχώρευσης, διότι πιέζει και ο χρόνος. Δύο λεπτά λοιπόν παρακαλώ ο καθένα και αναφέρομαι στου συναδέλφου. Η Σεσίλ Κέγγε τώρα, δύο λεπτά παρακαλώ, Σεσίλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Κλοντ, να ευχαριστήσω και τους εισηγητές μας, τους παρεμβαίνοντας για τα όσα είπαν. Θεωρώ ότι τα θέματα τα οποία επέλεξαν και μας παρουσίασαν πραγματικά θα πρέπει να μα απασχολήσουν πολύ γιατί συμφωνούμε, θεωρώ, με πάρα πολλά από τα σημεία τα οποία έχουμε καλύψει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ στους ανήλικους, στο μείζον συμφέρον των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Εδώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε όλα τα ψηφίσματα τα οποία έχουμε καταθέσει, εφαρμόζουμε την αρχή αυτή του μείζωνος συμφέροντος του παιδιού παντού. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο είναι οριζόντιο, μια προτεραιότητα προκαταρκτική. Αναφερόμενη στα όσα μας είπε η κυρία Τζαμφάνια για τους ασυνόδευτους ανήλικους, πραγματικά συμφωνώ ότι θα πρέπει εδώ πέρα να αφαιρθούμε και στην νομοθεσία Τζάμπα, μια νομοθεσία η οποία είναι αρκετά καινοτόμα, ακόμα και σε σχέση με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια Ιταλική νομοθεσία η οποία προβλέπει πολλές θετικές ρήτρες όσον αφορά την ένταξη των ανήλικων μεταναστών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να εμπνευστούμε από την νομοθεσία αυτή. Και η νομοθεσία αυτή προβλέπει και τον ρόλο του μέντορα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε και με το ζήτημα αυτό και με το ζήτημα των δικαιωμάτων. Δικαιώματα τα οποία όπως ισχύουν ακριβώς για τους ενήλικες θα πρέπει να ισχύουν, ισχύουν και για τους ανήλικες για τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα, την μπλε κάρτα. Και εδώ πέρα πάλι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η μεταφορά των δικαιωμάτων. Δεν φεύγει κάποιο από το σπίτι του αφήνοντα πίσω τα δικαιώματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα μεταφορά των δικαιωμάτων για όσου εγκαταλείπουν τη χώρα του. Επομένω, η πρόταση η οποία έγινε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ακριβώ επειδή θα ενισχύσει, πιστεύω, την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Σα ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ, για τώρα ο κύριος Βαλέρα. Uh, Κυρία Βαλέβα. Να σας ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα. Νομίζω ότι είναι θετικό αυτό που αναφέρατε για την υποτροφία. Αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλες τις χώρες, γιατί τώρα Κάποιες χώρες υποδέχονται, δέχονται τέλος πάντων τους αστυνομικούς ανηλίκους και κάποιες όχι. Στη Σουηδία πάντως ενσωματώνονται γρήγορα και μαθαίνουν τη γλώσσα. Αλλά πάντως είναι δύσκολο το τι θα κάνουν στα 18 γιατί υπάρχει ένα κατόφλι για την παιδεία. Τι είναι αυτό που το Τους χρειαζόμαστε και αυτοί χρειάζονται την παιδεία. Είτε μείνουν εδώ, είτε γυρίσουν πίσω. Τόσο αφορά το δικαίωμα στο παιχνίδι. Ε, βέβαια έτσι είναι σε μια οικογένεια, αλλά το πιο σημαντικό για αυτά τα παιδιά είναι να έρθουν κάποια στιγμή σύντομα μετά το δικό τους εργόμο οι γονείς τους είμαι το 86 ως δικηγόρος και ως ε, ερμηνείας ασχοληθεί και ήταν τότε πολύ πιο εύκολο να έρθουν ε, στη Σουηδία ακόμα και οι παππούδες τους. Μπορούσε κάποιος λοιπόν να κάνει το σχετικό αίτημα και το αίτημα μπορούσε να ικανοποιηθεί. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλουσί... Να από μια οικογένεια και ακόμα πιο σημαντικό να έχει τη δική του οικογένεια. Αυτά λέμε στη Σουηδία. Έχουμε και την μπλε κάρτα και πολλά χρόνια την χρησιμοποιούμε. Κόλλησε το θέμα στο Συμβούλιο. Ο πρόεδρος μας είναι ο εισηγητής για την έκθεση αυτή. Πάντως αυτό που προσπαθώ είναι να προωθήσω αυτή τη δική μας ειδική πρόταση για την ομοθεσία μας που ανέγεται στο 2008. Και είναι πολύ ευρία η αντίληψή μας και για αυτούς που έχουν πολύ ανεπτυγμένες δεξιότητες αλλά και για τους υπόλοιπους. Όλους, όλους τους χρειαζόμαστε να μας έρθουν. Και δεν έχουμε κάποιο μισολογικό κατόφλι. Τα συνδικάτα φυσικά έχουν όρια ε, για τους μισθούς και τις ανιδές κάθε κλάδο. Αυτά τόσο δεν είπα ότι πετύχαμε το τέλειο. Τόσο θα σας τα εξηγήσω και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπόντι, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο Λούκας και η Ρέιτσελ μπορούν να απαντήσουν στους βουλευτές που σχολίασαν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε βουλευτές, για όσα είπατε. Ας ξεκινήσω από την τελευταία παρέμβαση. Για αυτά που είπε η κυρία Βαλέρο, σας ευχαριστώ που μας είπατε τα της δικής σας εμπειρίας. Ναι, ναι, και εγώ επίσης ε, εργάζομαι με τους μετανάστες και ως δερμηνέας και ως ασκούμενη δικηγόρος. Ναι, ναι, το, είναι τέλεια, τέλεια τα αποτυπώνει όλα το δίκαιο. Κυρία Κέγγια και εγώ η Ιταλίδα είμαι και όντως ε, αυτός ο νόμος αποτελεί μία ε, απόκριση σε όλα αυτά τα οποία εδώ ε, αναφέρονται στη διεθνή σκηνή γενικότερα. Το πρόβλημα είναι, πρέπει να το τονίζουμε, ότι, είναι, ότι de facto έχουμε κάποιες μικρές κοινότητες παντού και όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο τέλο πάντων ή το κοινοτικό δίκαιο δεν τηρούνται για τα ασυνόδευτα παιδιά. Θέμα τι κάνουν οι κοινότητες. Αυτό είναι που μετράει. Και τι γίνεται με την ε, ε, πλαισίωση των παιδιών αυτών από κάποιες οικογένειες. Ε, βέβαια, το, καλύτερο για το παιδί είναι να έχει τη δική του οικογένεια. Παρά το να πηγαίνει σε κάποια οικογένεια, γερμανική, σουηδική, ιταλική κλπ. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Στην Ιταλία έχω μιλήσει στη δική μου πόλη καταγωγή μου με πολλούς μετανάστες, πολλά από αυτά τα παιδιά και τελικά ένα ένας 15χρονος πάει στο σχολείο από του 18 ανηλίκους που βρίσκονται στην πατρίδα μου. Και ένα ε, άλλο παιδάκι ήταν 8. Καλά, εντάξει, μου πήγανε σε ένα σχολείο. Αλλά τι γίνεται με τα παιδιά που είναι 17 γιατί λένε στις κοινότητε της πόλης ότι δεν ενδιαφέρονται οι μετανάστες. Είναι 17, θα ενηλικηθούν σε ένα χρόνο, δεν τους ενδιαφέρει το σχολείο. Γιατί είναι να βάλουμε αυτά τα παιδιά σε τελικά σχολεία. Ας τους βάλουμε στα τσιπία, δηλαδή στα σχολεία για εργαζόμενους και ενήλικες. Οπότε ε, αυτοί οι μετανάστες 15 με 18 αλλά και άλλοι νέοι μετανάστες από 18 και πάνω πάνε σε τέτοια σχολεία για 2-4 ε, ώρες τη βδομάδα. Τη βδομάδα. Τι να σας πω, ε, ίσως θα πρέπει να ψάξω και παραπέρα, αλλά η δική μου εμπειρία αυτά λέει. Λούκας, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για την ε, πρώτη δήλωση. Ε, θεωρώ ότι... Ε, εντάξει, η έρευνα είναι μια πάρα πολύ καλή διαξόδο, αλλά δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε σπουδάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλει να παραμείνει εδώ ή θα προχωρήσει στην έρευνα. Το άλλο είναι ότι χρειαζόμαστε και τα δύο, συμφωνώ πλήρω. Και αυτό θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα να ξεκινήσουμε με τους προσοντούχους. το κατοπίο δεν θα προκαλεί και αντιδράσεις. Και επίσης λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτό το θέμα είναι και μια προσωπική ιστορία. Το άτομο το οποίο έγραψε αυτήν την ιδέα είχε πει ότι ήθελε να πάει στη Γαλλία, είναι πολύ καλή φοιτήτρια κτλ. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να βρει δουλειά αφού τελειώσει νομική. Και όταν άρχισα να το σκέφτομαι, ε, γνωρίζω σχεδόν ένα άτομο με το ίδιο βιογραφικό στην Αυστρία, επίσης φοιτήτρια της νομικής, ε, δουλεύει για ΜΚΟ με πρόσφυγες ε, και φοβόταν ότι θα απελαθεί γιατί η αυστριακή κυβέρνηση άρχισε να σκέφτεται πως θα έπρεπε παραμένει νόμιμα στη χώρα κτλ. Οπότε το να το κάνουμε μόνο για τους ερευνητές ε, είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά ένα πρώτο βήμα μόνο. Δεν νομίζω ότι... Ε, ε, θεωρώ ότι όλοι όσοι αποφυτίσουν από εδώ θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι που πρέπει να αναφέρουμε, γιατί αναφέρατε την μπλε κάρτα. Ε, και την κυρία μου απασχολεί αυτό το θέμα. Ε, είμαστε πολιτικά περιορισμένοι όσον αφορά τα μέτρα της νόμιμης ε, μετανάστευσης και μετά υπάρχουν και πιο τεχνικές πτυχές γιατί είναι θέμα κυριαρχίας των κρατών μελών οπότε ένα τομέα που δεν έχει αναπτυχθεί λόγω αυτών των προβλημάτων. Παρόλα αυτά δεν ξέρω αν θέλουν οι βουλευτές θα μπορέσουν να επανέλθουν. Οπότε άτομα όπως η κυρία Βίξτρομ και οι άλλοι το γνωρίζουν ότι παρόλα αυτά καταφέραμε να περάσουμε κάποια μέτρα νόμιμης ε, μετανάστευσης. Οπότε αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Οπότε έχετε δικαίως ε, χαρακτηρίσει την ε, μπλε κάρτα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τους δύο. Τώρα θα περάσουμε στην Σιμών, στον Σιμών ε, για να μας παρουσιάσει τις δύο ιδέες του για να καταπολεμήσουμε τον αποκλεισμό των ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων. Λούκας θα παρουσιάσει και ιδέες για ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Σιμών, λοιπόν, προχώρα. Ευχαριστώ. Η πρώτη ιδέα που θέλω να παρουσιάσω έχει να κάνει με τον αποκλεισμό και τους νέους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε δίκτυα εξτρεμισμού, εγκληματικότητος και βίας. Οι νέοι θα πρέπει να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Στόχος βασική ιδέα είναι να καταφέρουμε να επανεντάξουμε στην κοινωνία του πιο αποκλεισμένου από την κοινωνία. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να πάρει έπειτα τη μορφή σχεδίου δράση που θα μπορούν να εφαρμόσουν οι τοπικέ κυβερνήσει παντού στην Ευρώπη. Ποια είναι η ιδέα αυτή καθεαυτή. Αν θέλουμε να μειώσουμε τη βία πρέπει να δούμε το όλο πλαίσιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που μπορούν να σπρώξουν ένα νέο, ναι, ένα νέο αυτό το καταστροφικό περιβάλλον. Θεωρώ, λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και το γενικό συνέστημα του κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε ομάδες κατά της δημοκρατίας και κατά των νόμων αν οι νέοι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να διαμορφώσουν εκ νέου τη ζωή τους και ότι μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία, τότε οι παράγοντες που τους έχουν κρατήσει εκτός κοινωνίας και εκτός του νόμου θα εξασθενήσουν. Πρόκειται λοιπόν για μια στρατηγική που θα επιτρέψει στους νέους να εγκαταλείψουν τον εξτρεμισμό καθώς επίσης και την εγκληματικότητα. Και θα ακολουθούν διάφορα στέδια εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συναντήσουμε τους νέους σε αυτές τις ομάδες στόχου. Μην περιμένετε να έρθουν αυτοί σε εσά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάτε να τους βρείτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κεντρίσετε το ενδιαφέρον του με ζητήματα που του ενδιαφέρουν, όπω οι πολεμικέ τέχνε για παράδειγμα. Δεύτερον, θα πρέπει να δημιουργήσετε την απαραίτητη εμπιστοσύνη προκειμένου οι νέοι από τις πληγήσεις αυτές κοινωνίες, περιοχές να αναλάβουν ένα πιο ηγετικό ρόλο, να ασχοληθούν περισσότερο με τα κοινά, να καταφέρουν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Εκεί πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Και τρίτον, η ομάδα αυτή στόχος θα πρέπει να ενταχθεί στη συνέχεια σε πολιτικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα στα Συμβούλια των Νέων. Έτσι λοιπόν οι νέοι συμμετέχοντες από τις πιο πληγήσεις περιοχές θα μπορέσουν πραγματικά να λειτουργήσουν ως μέντορες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να φέρουμε από κοντά νέου και τοπικέ κυβερνήσει, τοπική αυτοδιοίκηση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε του νέου και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποφεληθούν από τον νέο αυτό πόρο, του νέου δηλαδή. Αυτή ήταν η πρώτη μου ιδέα, τώρα θα περάσω στη δεύτερη. Η δεύτερη ιδέα έχει να κάνει με την προσωπική μου εμπειρία από τον τομέα της απαγκίστρωσης, απεμπλοκής των νέων από εξτρεμιστικές ομάδες και από εγκληματικές ομάδες. Έχω συμμετάσχει σε διάφορες ε, τέτοιες ε, ε, δοκιμές που γίνανε προκειμένου να καταφέρουμε να απομπλέξουμε τους νέους από τις ομάδες αυτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε νέα προγράμματα ενίσχυσης των νέων αυτών. Ποιο είναι το όλο υπόβαθρο τώρα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα αποδέσμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν στεφθεί με επιτυχία. Τα πιο επιτυχία από τα προγράμματα αυτά είναι αυτά που χρησιμοποιούν τους λεγόμενους formers στα αγγλικά, δηλαδή τους ε, ε, πρώην, ε, αν θέλετε, συμμετέχοντες σε εγκληματικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτοί να λειτουργήσουν ως μέντορες, ως καθοδηγητές. Είναι πολύ δύσκολο όμως να καταφέρουμε να εντοπίσουμε πραγματικά ποιοι είναι οι πρώοι συμμετέχοντες σε εγκληματικές αυτές ομάδες και δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστα είναι τα άτομα αυτά. Ενδεχομένω ο πρώην αυτό συμμετέχον σε εγκληματική ομάδα να μην έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να καταφέρει να νουθετήσει άλλου νέου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να πλαισιώσουμε του εκπαιδευτέ αυτού και να καταφέρουμε πρώτα βέβαια να του εντοπίσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα προγράμματα αυτά αποδέσμευση. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει μια δεξαμενή πόρων, ένα αποθετήριο αν θέλετε, με τα ονόματα των πρώην αυτών μελών εγκληματικών ή εξτρεμιστικών ομάδων, προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε του ανθρώπου αυτού ω εκπαιδευτέ, ω μέντορε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε πλατφόρμε με του νέου αυτοσυμβούλου για την καταπολέμηση τη ρίζοσπαστικοποίηση. Το δίκτυο RAN, ευαισθητοποίηση για την ριζοσπαστικοποίηση, μπορεί να μα παράσχει την πυρογνωμοσύνη του, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να μα παράσχει συγκεκριμένου διδάσκοντε, πρώην μέλη δηλαδή εγκληματικών ομάδων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρει να δημιουργηθεί το νέο αυτό μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε του ανθρώπου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μα δώσει απαραίτητου πόρου, προκειμένου να κλείσει το κενό αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Um, Τώρα και για του δύο που μα παρουσίασαν τι ε, θέσει του, αν έχουμε κάτι να απαντήσουμε. Κύριε να σα τα πω στα γερμανικά, λέει η κυρία Ζήμπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για το ότι αναφερθήκατε ε, στο θέμα της ε, πρόληψης και της ένταξης, ε, δηλαδή όταν οι νέοι, ειδικά οι νέοι, δεν αισθάνονται κομμάτι της κοινωνίας, και δεν υπάρχει κάποια ευκαιρία για να υπερευσιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό έχει διαφορές αρνητικές συνέπειες, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, ούτε καν για την εκπαίδευσή τους, αλλά πράγματι μπορεί να καταλήξει σε βία και εγκληματικότητα. Έχουμε αναφερθεί στις αθλητικές δραστηριότητες για μια πρώτη δυνατότητα επαφής και νομίζω ότι είναι μια σημαντική πτυχή. Στην ε, πόλη μου λένε ότι πρέπει να πάμε να τους βρούμε εκεί όπου βρίσκονται. Το θέμα λοιπόν της Βουλής των Εφήβων είναι ένα θέμα το οποίο ήδη έχει δοκιμαστεί σε πολλές πόλεις και δήμους της Γερμανίας για μένα σημαντικό είναι να υπάρξει μια διαδικασία για όλα τα κοινοβούλια που να διασφαλίζει ότι θα υπάρχουν ε, πολλοί και διάφοροι νέοι μετανάστες και μη, πλούσιοι και φτωχοί, ένα πολύχρωμο μείγμα νέων με διαφορετικά επιχειρήματα και επιθυμίες για καλύτερη ένταξη. Επίσης τα πράγματα αυτά αποχώρησης από αυτόν τον ε, χώρο είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα προγράμματα mentoring ε, τα οποία αναφέρεται. Υπάρχουν πολλά πετυχημένα μοντέλα γιατί βεβαίω κάποιος εμπιστεύεται κάποιον ο οποίος έχει περάσει την ίδια εμπειρία και μπορεί να του πει γιατί ήταν κακή η ιδέα η ριζοσπαστικοποίηση, ποιε είναι οι δυνατότητες για να ξεφύγει από αυτό. Υπάρχουν όντως κάποια προγράμματα αλλά σημαντικό είναι ακριβώς να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες που έχουμε με αυτά τα προγράμματα και πιθανώς να υπάρχει ναι. κάποια οικονομική στήριξη. Να κάνω τώρα μια μικρή παρατήρηση αν μου επιτρέπετε. Καλό θα ήταν τα κράτη-μέλη να μην τσακώνονται για κάθε ευρώ που δίνουν στον κοινοτικό προπολισμό. Όποιος θέλει ισχυρότερη Ευρώπη που θα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα θα πρέπει ακριβώς να δώσει και τους οικονομικούς πόρους. Σας ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Κρίσμπεκ. Σε ευχαριστώ, Κλοντ. Με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω για όλη αυτή την ευφυή, υπέροχη δουλειά για αυτό το πρόγραμμα. Μα αυτό θα πρέπει να γίνεται αυτή η ανταλλαγή εδώ στην Επιτροπή μας. Γιατί είναι διπλό το ενδιαφέρον όπως ε, τα είπαν και οι συνάδελφοι. Και έχουμε το Intergroup των Δικαιωμάτων των Ανηλίκων με συναδέλφους από όλες επιτροπές, οπότε και εκεί θα πρέπει να περάσουν όλα τα θέματα όσον αφορά για τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια, την προστασία αυτών των ανηλίκων και κυρίως τα θέματα για την Ευρώπη και αυτά που είμαι στην ε, εισαγωγή. Όλα αυτά το έχουν σχέση με την φύλαξη κράτηση τέλος πάντων των ανηλίκων ε, προσφύγων και την ένταξή τους. Τώρα όσον αφορά την ριζοσπαστικοποίηση, καταλαβαίνω το τι έχει προταθεί για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, για την επανένταξη των ε, βίων νέων, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ιδιορυθμίες που συντρέχουν ε, και τις άλλες προτάσεις για αυτό το θεματολόγιο σε σχέση με την οικοδόμηση σχέση εμπιστοσύνη, τόσο ώστε να σταματήσει ο καταστροφικός τρόπος ζωής που πολλές φορές ξεκινάνε αυτοί οι νέοι και που συχνά αυτό γίνεται χωρίς να το θέλουν ή χωρίς να το συνειδητοποιούν και αυτό να γίνεται μέσω αυτού του πουλου, όπως είπατε, αυτού του συστήματος ε, ε λειτουργιών στα πλαίσια και της Επιτροπής ε, της Αντιτρομοκρατικής. Το συζητήσαμε, ψηφίσαμε κάποια έκθεση και πέρα των άλλων θεμάτων που επεξεργαστήκαμε και συζητήσαμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της έκθεσης αφορά την ριζοφαστικοποίηση και την πρόληψη αυτής. Οπότε, ακριβώς με την έννοια των όσων και εσείς αναπτύξατε, προβλέπετε εκεί σε εισαγωγικά το πώς θα εκμεταλλευτούμε την εκμετάλλευση των παλαιότερα ριζοσπαστικοποιημένων ε, νέων που πια ξέφυγαν και αυτοί θα πρέπει να πάνε να μιλήσουν στους υπόλοιπους νέους για τους κινδύνους αυτής της ε, υπόθεσης. Οπότε, έτσι, τον έρχονται δηλαδή οι νέοι σε επαφή με τους υπόλοιπους ε, νέους, αυτό θα είναι ένα όπλο αντιμετώπιση. όπως τα είπατε. Αυτό που λέγατε για αυτή την ομάδα των ε, εκπαιδευτών ούτως υπήν. Έτσι θα καλύψουμε το θέμα του πόσο ευάλωτοι είναι οι νέοι. Έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε την πρόληψη της ριζοβαστικοποίησης. Α, κάτι που δεν άκουσα, αλλά αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη στο μέλλον. Όλη την προβληματική πρέπει να υπάρχει για ε, την ριζοβαστικοποίηση ε, μέσω του ίντερνετ. Καλά. Και διμερό μπορούμε να τα πούμε, εάν συμφωνείτε. Και πάλι ευχαριστούμε, μπράβο για την ποιοτική δουλειά σας και για αυτή την ε, ε, σημερινή ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστούμε πολύ, Σιμών. Θέλετε να απαντήσετε. Θέλετε να απαντήσετε στις παρατηρήσεις που ακούσατε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα θερετικά σας σχόλια να απαντήσω καταρχάς στην πρώτη παρέμβαση από την κυρία Σίπελ. Αναφερθήκατε, θίξατε πολλά από τα σημεία τα οποία ανέφερα και εγώ. Είπατε ότι όντω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τομέα του αθλητισμού για να έρθουμε σε επαφή περισσότερο με του νέου αυτού. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ επίση και σε αυτό που είπατε για την Βουλή των Εφήβων. Ενδεχομένω να μην ήμουν απόλυτα σαφή όταν παρουσίασαμε στα δύο αυτά λεπτά τι ιδέε μου. Ο δικό μου στόχο ήταν να ευαισθητοποιήσουμε και τους νέους αυτούς οι οποίοι δεν συμμετέχουν εξ ορισμού στην Βουλή των Εφήβων. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, νέοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πολιτική και που αυτόματα και φυσιολογικά θα συμμετείχαν σε μια βουλή των εφήβων, εγώ θέλω περισσότερο να καλύψουμε του νέου εκείνου οι οποίοι δεν θα πήγαιναν αυτόματα και εντελώ φυσιολογικά να συμμετάσχουν σε μια βουλή των εφήβων. Σε αυτού ακριβώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε από τους νέους αυτούς να αντλήσουμε τις λύσεις, γιατί ακριβώς οι νέοι αυτοί σε καθημερινή βάση βρίσκονται σε επαφή με φαινόμενα βίας, με ριζοσπαστικοποίηση, με εξτρεμισμό. Αν τους δώσουμε λοιπόν τους απαραίτητους πόρους, αν τους πείσουμε ότι όντως μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν και να αλλάξουν τα πράγματα, τότε οι ίδιοι μόνοι τους θα γίνουν φορείς των βέλτιστων αυτών πρακτικών. Και να κάνω ένα ακόμα σχόλιο για την κυρία που φοράει μαύρα. Δυστυχώ δεν θυμάμαι το όνομά σα. Είπατε ότι όντω θα πρέπει να υποφεληθούμε από τους νέους αυτούς που έχουν αυτή τη σχετική εμπειρία ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο στη δυνατότητα αυτή, να τα εκμεταλλευτούμε ακόμα περισσότερο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Και αν όντω εργαστούμε κατά αυτόν τον τρόπο, στον τομέα αυτό, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ω προ τον έλεγχο ασφάλεια, αν θέλετε, και να μπορούμε τελικά να δούμε πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε του νέου αυτού. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μεταμαύρη είναι η κυρία Ναταλή Γκρίσμπεκ, λέει ο πρόεδρο. Ποτέ δεν την έχουμε αποκαλεί στο παρελθόν, φαντάζομαι, γυναίκα με τα μαύρα, έτσι δεν είναι. Λούκα, ενδεχομένω να έπαιρνε το λόγο και για ένα λεπτό όσον αφορά του ανθρωπιστικού διαδρόμου. Δύο λεπτά, πολύ ωραία, δύο λεπτά. Μπορεί να μιλήσει για δύο λεπτά για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι δεν αφιλεγόμενα ζητήματα η ριοσπαστικοποίηση και η μετανάστευση σε διαβεβαιώ ότι είναι και τα δύο. Εκτός μικροφώνου παρατηρήσεις. Πόσο χρειάζεσαι, δύο ή τρία λεπτά. Δύο λεπτά Πολύ ωραία. Και Σεσίλια, εν συνεχεία μπορείς εσύ να πάρεις το λόγο και να αντιδράσεις τα όσα θα πει ο Λούκας. Σεσίλια Βίκστρομ, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια δυνατόν και εγώ. Πρόεδρο, ναι, αφού ολοκληρώσει ο τελευταίο ομιλητή, θα ακούσουμε πρώτα μία παρέμβαση όσον αφορά του ανθρωπιστικού διαδρόμου και μετά μπορείτε να πάρετε το λόγο, κυρία Βίξτρομ ή οποιοδήποτε άλλο, για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα. Okay. Yeah, of course. That's the one minute would be But I start. Okay, thank you. Okay. <laughs> thank you. Και το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να αναφερθώ και στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους πρόσφυγες. Πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά ο τόπος όπου υποβάλλονται αιτήσει για άσυλο, όχι στα κράτη-μέλη όπως γίνεται τώρα, αλλά στις πρεσβείες, στις προξενικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντού αλλού στον κόσμο. Θα γίνεται εκεί μια πρώτη συνέντευξη και θα γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση από τους ε, εργαζόμενους στην πρεσβεία ή το προξενείο για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Σύμβασης της Γενέβης. Εν συνεχεία θα λαμβάνει η απόφαση για το αν ο ετών μπορεί να πάρει το καθεστώς του πρόσφυγα ή όχι. Θεωρώ και ότι πάλι η λύση εδώ πέρα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, πρέπει να συμμετέχουν όλες οι χώρες. Η στρατηγική σύμφωνα με την οποία δεν θέλουμε κανέναν πρόσφυγα, ενδεχομένως να είναι δημοφιλής για κάποιους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ρεαλιστική. Γιατί αυτοί που φοβούνται ότι θα σκοτωθούν, ότι θα χάσουν τη ζωή τους, πάντα θα φεύγουν από την εμπόλεμη χώρα στην οποία ζουν. Υπάρχουν πολλές φορές και πρόσφυγε, οι οποίοι μολονότι ζουν και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε αντικσοότητε, δεν μπορούν να πάρουν το καθεστώ του πρόσφυγα σύμφωνα με την Σύμβαση τη Γενέβη. Αυτό συμβαίνει με όσου αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, τι δυσμενεί επιπτώσει των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε από τώρα, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολλού πρόσφυγε στο μέλλον εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και απαραίτητε τροποποιήσει στην Σύμβαση τη Γενέβη, προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε και αυτού του ανθρώπου. Επίση, μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι στι πρεσβείε Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτε χώρε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την κατάσταση που ισχύει στι χώρε αυτέ και μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν αν υφίστανται προποθέσει χορήγηση του καθεστώτο τη διεθνού προστασία. Ας μην ξεχνάμε ότι η αύξηση των ελέγχων σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σταματήσει τη δράση των διακινητών. Απλώς θα αυξήσει την τιμή που προτείνουν αυτοί οι διακινητές στους πρόσφυγες προκειμένου να τους περάσουν προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι η πρόταση αυτή που κάνω, προκειμένου δηλαδή να αξιολογούν οι αιτήσει ασύλου σε τρίτε μονοχώρε από τι προξενικέ αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια αρκετά τολμηρή πρόταση. Παρ' όλα αυτά, θα θέλω όμω και τη δική σα την αντίδραση. Η Σεσίλια, ναι, συμφωνώ πλήρω. Πράγματι, πρέπει η Ευρώπη να συνέλθει και να δράσει ενωμένη. Αυτή είναι η θέση αυτού του θεσμικού οργάνου. Δυστυχώ υπάρχει και ένα άλλο θεσμικό οργάνο που δεν έχει ξεκινήσει καν να ασχολείται με την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Μην κατηγορείτε λοιπόν εμάς. Εμείς είχαμε μια φανταστική θέση και εγώ είμαι ανά πάση στιγμή έτοιμη για διαπραγματεύσεις. Αυτά. Για αυτό. Να επανέλθω τώρα σε κάτι το οποίο αναφέρατε πριν ε, για τα παιδιά, μετανάστες και την κράτηση. Θεωρώ ότι έχει φτάσει η στιγμή να σταματήσει η κράτηση ανηλίκων ε, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όπως ε, καταφέραμε κάποτε να καταργήσουμε τη θανατική ποινή, τώρα έχει φτάσει η στιγμή να πούμε ότι πρέπει να δράσουμε ενωμένοι. Τέλο, η επανένωση των οικογενειών είναι ένα άλλο θέμα πολύ κρίσιμο και από αυτού τα κράτη-μέλη τώρα συμμετέχουν, όλα τους θα έλεγα, να κάνουν ό,τι μπορούν για να ανοίξουν τα χείρα τους και ακόμη και η χώρα μου η Σουηδία που τα έχει καταφέρει τόσο υπέροχα στην επανένωση των οικογενειών τώρα σχεδόν όλα τα κόμματα με κάποιες ε, εξαιρέσεις, το δικό μου κόμμα δηλαδή. Ακόμα και οι σοσιαλιστές, ε, το μεγάλο συντηρητικό κόμμα είναι κατά της κοινωνικής επανένωσης. Και μιλάμε για τον 21ο αιώνα, όπου έχουμε αυτή τη στιγμή φέτος ένα χαμηλό ιστορικό εισόδου μεταναστών θυμάμαι μια αμερικανική παροιμία που είχε χρησιμοποιήσει και η Χίλαρη Κλίντον για το ότι όλο το χωριό μεγαλώνει το παιδί, απέχουμε πολύ από αυτό και τα παιδιά τους θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά στο μέλλον. Και τα παιδιά μας οπωσδήποτε. Αναγνωρίζω λοιπόν αυτά τα οποία λέτε και βεβαίως είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο αναφέρθηκε ότι έχουμε μια διακομματική ομάδα για τα παιδιά εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ και κυρία Μπεριγκίτ. Ε, θέλετε να πείτε κάτι. Θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στο αίτημα αυτό περί ανθρωπιστικής βίζας και να τονίσω ότι αυτό θα μας βοηθούσε σε πολλούς τομείς. Ε, πρώτα απ' όλα να σταματήσουν αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα που προσπαθούν να μπάσουν κόσμο να τους διαβεβαιώσουμε ότι μπορούν να μείνουν εκεί που είναι και θα έχουν ασφαλείς διόδους να ζητήσουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ας είμαστε ειλικρινεί. δεν με χαροποιεί αυτό και με την κατάσταση και η ανθρωπιστική βίζα δεν λένε ότι αυτά τα άτομα θα, έχουν, ε, θα λάβουν άσυλο, απλά θα μπορέσουν να φτάσουν ασφαλώς στην Ευρώπη για να εξεταστεί η αίτησή τους. Και λένε ότι αυτός θα είναι ένας παράγοντας που θα προσελκύει. Δεν είναι αλήθεια αυτό. μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων δεν έρχεται στην Ευρώπη και πρέπει να διευκολύνουμε αυτού που θέλουν να ζητήσουν βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πέρα συμφωνώ πλήρω μαζί σας. Δεν θα επικεντρωθούμε στο να χτίζουμε σύνορα και φράχτες. Αν ο κόσμος θέλει θα έρθει. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να διασφαλίσουμε ανθρωπιστικές βίζες, επανεγκατάσταση. Ε, σύντομα όμως, Μπριγκίτε, έτσι, σύντομα, σε παρακαλώ. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε αυτά και να πείσουμε, ελπίζω τα κράτη-μέλη, να δουν το θέμα της μεταγκατάστασης. Ελπίζουμε να επανέλθει η ανθρωπιστική βίζα. Ε, θα έχετε εσείς ε, τον τελευταίο λόγο λοιπόν. Θα ήθελα να μιλήσω στα γερμανικά, αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας άκουσαν. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ κρίμα ε, το ότι δεν υπάρχει κανένας αυστριακός ε, ευρωβουλευτής παρά το ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Το FPE θα έπρεπε να είναι εδώ γιατί τα τελευταία τέσσερα χρόνια μόνο για αυτό το θέμα μιλάνε. Επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρόντες ευρωβουλευτές ε, για τις δηλώσεις ε, που έκαναν. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι είχα την ευκαιρία να κάνω το γύρο της Αυστρίας ε, το καλοκαίρι. Μίλησα με τον κόσμο για το τι τους απασχολεί και στην Νόιστατ εκεί πέρα που είναι προπύργιο του ΕΦΠΕ σε μια πραγματικά εργατική συνοικία και αν μιλήσει κανείς δύο λεπτά τους ανθρώπους και ξεπεράσει το θέμα των προσφύγων, αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κακοί. Είναι άνθρωποι απογοητευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την επόμενη προεκλογική εκστρατεία. επικεντρωνόμαστε σε αυτό το θέμα γιατί τα άτομα αυτά απλά περιμένουν πραγματικές λύσεις για τα προβλήματά τους. Δηλαδή τους ζητάει απασχόληση, νίκη που συνεχώς ανεβαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από αυτά, γι' αυτό δεν ακούω τίποτα από την Ευρώπη. Αυτή είναι λοιπόν η παράκλησή μου. Ε, μακάρι να είχαμε χρόνο να ακούσουμε άλλον ένα γύρο από την ε, Ρέιτσελ και την Σιμών. Αλλά... Φανταζομαι και εσείς ε, ωραία θα τα λέγατε. βεβαίως αυτά τα ζητήματα μας απασχολούν στην Επιτροπή μας ε, και ακριβώ προσπαθούμε να ασχοληθούμε με συγκεκριμένες πτυχές αυτών των ζητημάτων. Και γεγονό είναι ότι οι βουλευτές οι οποίοι απάντησαν είναι βουλευτές οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα στο νομοθετικό μέτωπο ή μια συνάδελφος ασχολείται με τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου αυτό ακριβώς ε, κάναμε αυτή την εκδήλωση γνωρίζοντας ότι δεν θα έχουμε και πολλούς βουλευτές γιατί είμαστε αρκετά πολύ άσχολοι αλλά έπρεπε να ξεκινήσει ο διάλογος ε, με εσάς ε, και με τους υπόλοιπους εντός του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και τους ε, καλεσμένους μας ε, και όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Και αυτός ε, μετά του tweet και πέρα γράφει ωραία πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήρθαν και απάντησαν. Και βεβαίως μιλάμε για πραγματικά νομοθετικά ζητήματα τα οποία εξελίσσονται. Και τώρα θα συνεχίσουμε τη συνεδρία με κάποια από τα ζητήματα αυτά τα οποία αναφέρατε και ελπίζω στην επόμενη θητεία να δούμε πώς θα πάνε αυτά τα ζητήματα της μετανάστευσης, της ε, ρίζος παστικοποίησης κτλ. Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστώ προσωπικά και τους ε, τρεις. kind of really boring end to this when I have to go into another agenda. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Οπότε συμπαθάτε μας για την διασύνη. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, colleagues, we can go on. Προχωρούμε, συνάδελφοι, στο σημείο παριθμών 4. Αργήσαμε λίγο. Um, so we go now to the... Και οπότε προχωρούμε τώρα στο πρόγραμμα για δικαιώματα και αξίες. Η Μπόντιλ είναι εδώ που είναι κάτι το θετικό και τώρα αρχίσουμε την ανταλλήγη των απόψεων σαν αφορά τις ε, που έχουν κατευθεί για αυτό το πρόγραμμα της 2021 21 21-27 που γνωρίζετε εδώ πέρα έχουμε τους στόχους για το πρόγραμμα για τον προϋπολογισμό 21-27 και έτσι ανεφάλου προχωρούμε μια που έχουμε καθυστερήσει ε, προχωρούμε και δίνουμε τον λόγο στην ε, εισηγήτρια Μπόντιλ Ευχαριστώ πολύ βάλτε τα ακουστικά σας και πρώτα όλα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες εισηγητές. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία στα πλαίσια της δουλειάς της Επιτροπής μας. Να ευχαριστήσω πάντως και την ε, συνεισηγήτρια αλλά επίσης ε, και τους συναδέλφους από την Πολιτική Επιτροπή και την Επιτροπή Γυναικών, αλλά ΑΦΚΟ και, και, άλλες, και άλλες, γιατί τελικά ήμασταν πάρα πολύ συναρμόδιοι για αυτό το πρόγραμμα, για αυτή την έκθεση που αφορά δικαιώματα και Οπότε μέχρι τώρα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά κατά τη συνεργασία μας. Όταν αναλάβαμε αυτό το θέμα, το συζητήσαμε και ε, είχαμε το θέμα της συνέχισης ε, του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεύρυνση της συνεργασίας. Όσον αφορά τους φορείς, τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018. Αλλά το θέμα είναι ότι πέραν της αύξησης της πρικοδότησης του προϋπολογισμού είπαμε ότι θα έπρεπε να καλύψουμε περισσότερα θέματα, θα έπρεπε να καλύψουμε περισσότερους τομείς. Όμως επειδή έγιναν οι περικοπές δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων θα πρέπει να τα καταφέρουμε με όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκονται τα πράγματα, έχουμε ένα σωρό τροπολογίες, πολλέ από αυτές κινούνται στο ίδιο μήκος κύματο. Τέλο πάντων ε, υπάρχει συνένεση ευρεία στα περισσότερα σημεία. Ήδη με τους κοιόδης ηγητές έγινε μια συνεδρίαση ε, Είχαμε συμβαστικές τροπολογίες. Για τα πιο δύσκολα πάντως υπήρχε συνένεση. Θα τα ξαναπούμε και ελπίζω ότι θα βρεθούν λύσεις όπου χρειάζεται. Έχουμε τους βασικούς στόχους. Δεν θα πρέπει να θυγούν τα υπάρχοντα προγράμματα. Βέβαια, χρειάζονται περικοδότηση αλλά πάντως το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια συνένεση για το πρόγραμμα γενικώ. Και κάποια άλλα ζητήματα πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε το και το ψήφισμα του Απριλίου του 18, οπότε θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαδρομή και έχουμε τη, το, τον, τον πυλώνα της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε κάποια σχέδια, προγράμματα σε επίπεδο εθνικό και τοπικό. Έχουμε την εμπλοκή ε, της κοινωνίας των πολιτών, κάποιων ε, οργανώσεων και οργανισμών ε, καταπολέμηση της διαφθοράς, θωράκηση της προστασίας των δικαιωμάτων. Αυτά όλα είναι αλλά υπάρχει και άλλη μια πρόταση, ότι δηλαδή θα ήταν πιο εύκολο για τους μικρού σχετικά οργανισμού και οργανώσει να μπορούν να ζητήσουν μέσω του προγράμματος ε, πληκοδότηση και έτσι να διευκολυνθεί η δουλειά τους, να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή, να υπάρχει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την συναπόφαση για την αξιολόγηση του προγράμματος. Έχουμε τρία βασικά ζητήματα, επομένω που προέκυψαν και οι συνάδελφοι μπορεί να έχουν και κάποια άλλα ζητήματα αναδείξει. Η ψήφιση θα γίνει στις 10-12 ε, στην Επιτροπή και τον Ιανουάριο θα αρχίσει ο τριμερής διάλογος. Ελπίζω. Ελπίζω ότι πριν λήξει εντολή θα έχει κλείσει το θέμα. Άρα θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνάντηση με τους πιο ηγητές. Έχουμε και κάποια ζητήματα που εγκρεμούν, κάπως πιο δύσκολα από τα άλλα, αλλά ελπίζω ότι εκεί θα τα διεκπαιρεώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Μποντιλ. Όντω, έχετε καταβάλει πολλέ προσπάθειε και μπλέκονται και πολλοί σκιώδει εισηγητέ, καθώ επίση και εισηγητέ από συνδεδεμένε επιτροπέ. Ορισμένοι είναι παρόντε εδώ σήμερα. Α του ακούσουμε και ξεκινάμε με τον Μιχάλ Μπόνι, εξ ονόματο του ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ πολύ. όντω πολλέ φορέ συζητήσαμε το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι είναι από, από τις πιο σημαντικέ λύσεις που θα μπορούσε να προτείνει και να προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για προπολογισμό και όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νέο προπολογισμό και νομίζω ότι ο νέος αυτός προπολογισμός αποτελεί αν θέλετε κοινό αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών όλων των πολιτικών ομάδων καταφέραμε να τριπλασιάσουμε τον προτινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προπολογισμό και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό τώρα είναι να καταφέρουμε ε, να διατηρήσουμε ξεχωριστά τα σκέλη αυτά που μας παρουσίασε η Μπόντιλ και ιδίω να κρατήσουμε ξεχωριστή τη χρηματοδότηση για το σκέλος των αξιών. Και υπάρχει και σύγκληση μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών ομάδων όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος Δικαιώματα και Αξίες. Να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια που κατάφερε να προετοιμάσει μια πολύ ισχυρή πρόταση που θα αποτελέσει μια πολύ σταθερή βάση μελλοντικών διαπραγματεύσεων μεταξύ εισηγητών και σκιωδών εισηγητών και συμφωνούμε από κοινού ότι θα πρέπει προφανώ να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, να προωθήσουμε περισσότερο τα όσα λέγονται στο άρθρο 2 τη συνθήκη για τι αρχές και τις αξίες. Και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σκέλος, το σκέλος αξίες της Ένωσης και να επικεντρωθούμε περισσότερο επίσης στις ομάδες εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και κυρίως σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στις διάφορες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και νομίζω ότι προβλέπονται και διάφορες λύσεις φιλικές προς τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, να καταφέρουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία που πολύ συχνά βαραίνει τις οργανώσεις αυτές. Συζητήσαμε επίσης όλε τι πτυχές του προβλήματος αυτού, τη λειτουργία του δηλαδή, το μοντέλο το οργανωτικό το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί, το πώς θα καταφέρουμε να στηρίξουμε οργανισμούς σε τοπικό επίπεδο. Ενδεχομένως να προτείνετε μερικές φορές από εμά μια διαφορετική διατύπωση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα δικαιώμα, δικαιωμάτων και αξιών ως ένα θετικό πρόγραμμα επαναξιολόγησης των αξιών μας. Δεν στρεφόμαστε κατά συγκεκριμένου κράτους μέλους. Σε καμία περίπτωση θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε κανέναν. Και είμαι κατά του να γίνεται μία στη γενικότερη αυτή συζήτηση που έχει να κάνει με την μη εφαρμογή του κράτους δικαίου ή την αιρεσιμότητα που μπορεί να προκύπτει από τις αδυναμίες εφαρμογής του κράτους δικαίου. Νομίζω ότι η προτινόμενη λύση θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Ευελπιστώ ότι θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω από το Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να έχουμε εμεί μία λύση η οποία να μπορεί να λειτουργεί αλλού, αλλά μία λύση η οποία να μπορεί να λειτουργεί ρεαλιστικά εδώ για τα κράτη-μέλη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε αν ορισμένες λύσεις προτείνονται για το κράτος δικαίου, εν γέννη και θεωρητικά συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενταχθούν στην πρόταση αυτή και να φέρουμε εδώ πέρα στην αιρεσιμότητα, δηλαδή το να περιοριστεί ή να διακοπεί η χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων σε συγκεκριμένε χώρε όπου παρατηρούνται προβλήματα με το κράτο δικαίου. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το μελετήσουμε λίγο περισσότερο γιατί το ζήτημα τη αιρεσιμότητα αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Όπω είπε και η Μπόντιν, πιστεύω ότι μέσω των συμβαστικών τροπολογιών θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή βάση που θα μας επιτρέψει στις 10 Δεκεμβρίου να εγκρίνουμε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη και εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η Σεσίλ και τώρα εξ ονόματος των Σοσιαλιστών, έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ, Κλοντ. Όπως είχα τη δυνατότητα να το πω και στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια όχι μόνο για την αξιέπαινη εργασία που έχει κάνει σε σχέση με τις τροπολογίες και όλες αυτές τις αλλαγές που επέφερε τελικά στο κείμενο αυτό, αλλά επειδή πραγματικά έλαβε υπόψη και τις συγκεκριμένε τροπολογίες μας. Ξέρω ότι ε, από τεχνικής ε, πλευράς ε, προσπαθεί γρήγορα αυτή τη στιγμή η συγγήτρια να ενσωματώσει όλες αυτές τις τροπολογίες. Ευελπιστώ λοιπόν ότι θα συμμετάσχουν ε, θετικά όλε οι πολιτικέ ομάδε για να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Όσον αφορά τώρα τι πιο λεπτομερεί τροπολογίε, τι οποίε καταθέσαμε εξ ονόματο ομάδα σοσιαλιστών, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθεια που κατέβαλε να τι ενσωματώσει, ιδίω στην καταπολέμηση κάθε μορφή μυσαλλοδοξία, είτε αυτή εμφανίζεται στο διαδίκτυο είτε εκτό διαδικτύου. Για μα αυτό αποτελούσε σαφή προτεραιότητα. Προφανώ εξακολουθώ και είμαι πάρα πολύ πεπισμένο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πρόγραμμα πρόγραμμα το οποίο να λαμβάνει υπόψη και την ε, αξία της ε, ισότητας καθώς επίσης και την ιδιότητα του πολίτη. Ας μην ξεχνάμε επίσης και το ζήτημα βέβαια της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Δύο ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, προφανώς είμαι υπέρ μια σημαντική αύξηση της προβλεπόμενης χρηματοδότησης. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλέ και μεγάλες και η ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών που καταπολεμά το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τη μυσαλλοδοξία, τη ρητορική μίσου, ε, καθώ επίση και τον βίο εξτρεμισμό, προφανώ χρειάζεται μια έντονη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φέρει πέρα στο έργο τη. Να συγχαρώ για ακόμη μια φορά την εισηγήτρια, η οποία ακολούθησε τον οδικό χάρτη τον οποίο εμεί είχαμε προτείνει στην αρχή της όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή διευθετηθούν οι τεχνικές αυτές λεπτομέρειες. Μπορούμε να οριστικοποιήσουμε και να εγκρίνουμε το πρόγραμμα αυτό μέχρι το τέλος της δικής μας θητεία. Ευχαριστώ πολύ. Σίλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος του ECR τώρα ο κύριος Γιούρα και έχει το λόγο. Παρακαλώ. Bardzo E, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις ε, προηγούμενες ε, συζητήσεις μας ε, για το θέμα αυτό και για του Μίχαλ Μπόνι είχαμε παρουσιάσει την επιφυλακτικότητα μας για, πεν, για αυτούς τους μηχανισμούς και την αντικειμενική εφαρμογή τους. Οπότε έχουμε υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες για κάποιες εγγυήσεις ε, για αυτά τα οποία θα μπορούσε να εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά μια μονομερή προσέγγιση. Συγκεκριμένα επισημαίνουμε το άρθρο 17 της Συνθήκης ε, που μιλάει για συνεχή διάλογο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ε, κοινότητες και τις θρησκευτικέ αρχές. Επισημαίνουμε επίσης το θέμα των οικογενειακών οργανώσεων. Ε, γνωρίζουμε πως η τωρινή δημογραφική κρίση στην Ευρώπη σχετίζεται με την κρίση της οικογένειας ε, και θεωρούμε ότι η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα μπορούσε ακριβώ να επιβεβαιώσει τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί βασικών δικαιωμάτων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αξιολογηθεί στο έργο αυτό είναι να περιληφθούν οι τροπολογίες μας ε, στην αναζήτηση συμβαστικών προτάσεων. Δεν θα τις συζητήσω όλες, αλλά προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνουν οι προτάσεις μας. Και να δούμε επίσης πώς έχουν ε, οι εγγυήσει ε, για να δούμε με μεγαλύτερη πιστοσύνη τις ιδέες που αναφέρονται εδώ. Σας ευχαριστώ Σόφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί στηρίζουμε ολόψυχα την γραμμή του εισηγητή τον οποίο ευχαριστούμε για την επικοδομητική προσέγγιση. Μία πρόταση που θα θέλαμε να περιληφθεί εδώ είναι το 5% το αποθεματικό ανάγκης εκεί όπου υπάρχει προφανής παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση ενός κράτους μέλους. Ε, στην οποία περίπτωση πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει ένα αντίβαρο. Υπάρχει αυτό και σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. Και ίσως να υπάρξει κάτι το κατεπήγον και που να αφορά αυτά τα ζητήματα. Μετά, αντιδρώντας σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Μπόνι μόλις δεν θεωρώ ότι το μέσο αυτό στρέφεται ποτέ κατά κάποιου κράτους είναι υπέρ των πολιτών και στα κράτη εκείνα όπου η κυβέρνηση δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και στο δύσκολο στην κοινωνία των πολιτών, στους πολίτες της δηλαδή, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να ξεχάρισουμε το τι εννοούμε αιρεσιμότητα. Γιατί μόλις άκουσα τον Μίχελ Μπόνι να λέει κάτι για αιρεσιμότητα, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σχέση με το θέμα μας. Ε, αφορά τον προπολογισμό, είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Δεν με ενθουσιάζει, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει σε γενικέ γραμμές. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι θετικό το ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια είχε ένα τέτοιο μέσο στον προπολισμό εκτός της Ένωσης, αναγνώρισε επιτέλου ότι χρειάζεται ένα τέτοιο μέσο ε, για το εσωτερικό της Ένωσης, για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα υπερασπίσουν αυτούς. Έχουμε τα μέσα λοιπόν τώρα να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ Σοφή. Κάποιος άλλος. Ε, Μίχαλ. Μία κουβέντα Σοφή. Συμφωνούμε ότι πρέπει να προωθήσουμε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να διατηρήσουμε τη δημοκρατία, τις αξίες, το κράτος δικαίου, τον δημοκρατικό διάλογο και να είμαστε ανοιχτοί. Από την άλλη, πρέπει να μιλήσουμε και για κάποιες πρακτικές δυνατότητες. Και νομίζω θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό στις μεταξύ μας ε, συναντήσεις. Ναι, ναι, πολύ, πολύ δουλειά. Μπούντο. Ε, είναι για τις 10 Δεκεμβρίου. Θέλεις να μας πεις κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, εκκρεμούν κάποια ζητήματα με την οποία δεν έχουμε συμφωνήσει ανάμεσα στι πολιτικέ ομάδε, άρα και για αυτά θα πρέπει να βρούμε μια κοινή λύση. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την απαραίτητη πλειοψηφία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία τα προσεγγίζουμε διαφορετικά, άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά, να καταφέρουμε να συγκεράσουμε λίγο τι διστάμενε απόψει. Το θέμα δεν είναι ότι είναι κάποιο κατά τη μία η τη άλλη χώρα το οποίο θέλουμε να στοχευσουμε κατα μια χώρα. είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ότι θα τηρούν, θα προστατεύουν, θα προασπίσουν με τον ίδιο τρόπο τι αξίε και τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, αν σύμφωνα με το άρθρο 2 τη Συνθήκη ή σύμφωνα με άλλα άρθρα μια χώρα υπολείπεται του ευκταίου αυτού επίπεδου, θα πρέπει να έχουμε εμεί ένα μηχανισμό, ένα μοντέλο που θα μα επιτρέπει να φέρουμε τη χώρα αυτή στο σωστό δρόμο πάλι. Σε καμία περίπτωση όμως μέσω τη έκθεσης αυτή δεν στρεφόμαστε κατά της μία ή της άλλης χώρας. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much, and good luck. και εμεί ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη και καλή συνέχεια και να ευχαριστήσουμε και τους κοιόδης συγητές που συνεργάζονται για το ζήτημα αυτό με την Μπόντιλ. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, από κοινού τα σημεία 5 και 6. Έχουμε εδώ πέρα τη σύναψη συμφωνιών περί με την Αλβανία και με την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Μπόντιλ και πάλι είναι αρμόδια, η οποία δουλεύει πολύ σκληρά σήμερα. Έτσι δεν είναι. Μία ακόμα παρέμβαση από την Μπόντιλ σήμερα το πρωί. Το απόγευμα μάλλον. Λοιπόν, Μπόντιλ, σου ξαναδίνω το λόγο για τα ζητήματα αυτά. Παρακαλώ. I, I uh, suppose we talk about the both. Ε, και για τα δύο ζητήματα. Δεν είπατε. Ο πρόεδρος, αν δεν σε πειράζει, ναι, να τα συζητήσουμε από κοινού. Αυτό το, το καθεστώς σε σχέση με την Αλβανία, καθώς και τη συμφωνία με την πρώην γιουγκοσλαβική ε, Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σε πειράζει, μπορείς. Ωραία, ας τα πω στα σουηδικά λέει η κυρία η Και μαζί με τους ε, ε πρασίνους με το θέμα έχουν κριτική προσέγγιση όσον αφορά αυτές τις σχέσεις με τρίτες χώρες, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει κάτι να ρυθμιστεί και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μέσον η διαδικασία να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος, να υπάρξει εποπτεία και να υπάρξει κατανομή των ευθυνών, επιμερισμός των ευθυνών, πρώτα-πρώτα. Ε, έχουμε την Αλβανία, έχουμε μια σειρά συμφωνιών που έχουν συναφθεί πάρα πολύ σημαντικές. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει ένα καθαρό πλαίσιο των σχέσεων. Και με αυτές τις συμφωνίες να υπάρξει κατοχήρωση θημεριδών δικαιωμάτων, το δικαίωμα του ασύλου, να κατοχυρεθεί η αρχή της, ε, του σεβασμού της αξιοπρέπειας, το ε, δικαιώματα των ανηλίκων κλπ. Οπότε χρειάζεται και ένας λειτουργικός ε, μηχανισμός ενδίκων μέσων, κανόνες για το βόρος της αποδείξεως και να καλυφθεί και ο τομέας του ε, αστικού δικαίου αλλά και του ποινικού δικαίου και δικονομικά ζητήματα οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι όλα τα δικαιώματα, τα έγγραφα που χρειάζονται να τα λάβουμε υπόψη και για τις δύο αυτές ε, συμφωνίες θα πρέπει οι τροπολογίες να κατατεθούν μέχρι τις 28 Νοεμβρίου αλλά εν πάση τελικά πρόκειται για τη διαδικασία που λέμε ναι ή λέμε όχι. Άρα και οι τροπολογίε σε αυτό πρέπει να κατατείνουν ναι ή όχι. Άρα ε, ψηφοφορία στις 28 Νοεμβρίου στην Επιτροπή. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε ταυτόχρονα. Πάντως για την πήγαμε δελταμή δεν έχω ακόμα όλα τα στοιχεία, αλλά τέλος πάντων ε, ε, πρόκειται για το ίδιο σχήμα που ακολουθούμε και εν προκειμένου. Οπότε ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ό,τι χρειάζεται για να ψηφίσουμε τότε. Ο Πρόεδρος. Ωραία, Μπόντιλ, σε ευχαριστούμε. Οπότε, προθεσμία για τροπολογίες 28 Νοεμβρίου. Ναταλή, είσαι η μόνη παρούσα από τους και τις σκιώδεις εισηγητές. Ναι, ναι, δύο λόγια μόνο, σύντομα, Κλοντ. Έχουμε αυτές τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου για αυτή τη συμφωνία περί με την ε, Μακεδονία και την Αλβανία. Είμαι στο ίδιο με την ε, Μπόντιλ. Σημαντικέ οι συμφωνίε με αυτέ τι τρίτε χώρε. Και εγώ επίση θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η ρύθμιση να είναι σαφές. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για όλη την μέχρι τώρα δουλειά της. Α, κάτι το οποίο δεν ανέφερε η Μπόντιλα. Προφανώς όμως το γνωρίζει ότι η εν λόγω συμφωνίες λαμβάνουν υπόψη πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και ορίζουν ότι υπάρχει μια διαδικασία ε, άσκησης προσφυγής όπως ακριβώς ε, γινόταν και στο παρελθόν. Είμαι αισιόδηση εισηγητή για την πολιτική μου ομάδα όσον αφορά ε, την ε, Frontex. Αυτό θα το συζητήσουμε αύριο. Οπότε και είμαι σε θέση να γνωρίζω τις σχετικές διατάξεις. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μας για να υπάρξει όσο γίνεται περισσότερη ενημέρωση, πιο πολλά στοιχεία και έτσι τελικά να είμαστε ακριβείς και σαφείς σε ό,τι θα περιέχει αυτή η ρύθμιση και έτσι θα βοηθήσουμε την εύρυθμη εφαρμογή της συμφωνίας και κατά την εφαρμογή του να μπορεί να αξιολογείται η κατάσταση. Πολύ σημαντικό αυτό έτσι όπως έχει η σημερινή συγκυρία για τα εξωτερικά σύνορα και τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία Ναταλή. Σε ευχαριστούμε. Πολύ σημαντική και η διαδικασία και σε σχέση με συνοριοφυλακή και εκτοφυλακή. Δεν έχουμε τροπολογίες, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, μέχρι τις 28 δεκάτου, ό,τι γίνει. <laughs> That's fine. Thank you. Thank you very much. Και πάλι σας ευχαριστώ. ο πρόεδρος. Έχουμε τώρα το επόμενο θέμα, συνάδελφοι. Πάμε στο 7 και είναι αυτό το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο. Έχουμε εδώ 15 τροπολογίες. Η Κίνγκα είναι η εισηγήτρια. Εδώ είναι. Είναι η εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Να της δώσουμε το λόγο. 15 τροπολογίες, Κίνγκα. Πες μας. Ευχαριστώ πολύ, να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ηγητές για την επικοδομητική στάση που κράτησαν. Στην συνεδρία των σκιωδών εισηγητών χρειάστηκε να αποσαφηνίσουμε διάφορες πτυχές της πρότασης εγώ παρουσίασα την πρόταση αυτή και στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα για μία ακόμη φορά να τονίσω ότι η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ως στόχο να απλουστεύσει τις διατυπώσεις για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν χάσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και βρίσκονται σε τρίτη χώρα, στην οποία η χώρα τους δεν έχει πρεσβεία ή προξενική αρχή. Άρα απευθύνονται σε πρεσβεία ή προξενική αρχή άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βασικά του βοηθά, καλείται να του βοηθήσει να επιστρέψουν στι πατρίδε του. Δεν πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό, ήδη φύσταται από το 1996, αλλά έκτοτε, όπω ξέρετε, πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και τον υφιστάμενο μορφότυπό του ε, το έγγραφα αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη όλε τι προδιαγραφέ ασφαλεία που έχουν τα υπόλοιπα τα εξωτικά έγγραφα. Επομένω, δεν παράσχουν συγκεκριμένη προστασία όσον αφορά την απάτη, την παραποίηση. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν εκδίδουν πλέον αυτό το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ο μορφότυπος αυτού του εγγράφου. Και υπάρχει όμως και μια νομική υποχρέωση η απόφαση αυτή του 1996 δεν συνάδει με την οδηγία για την προξενική προστασία του 2015, άρα θα πρέπει να γίνει αυτή η ευθυγράμμιση. Ήδη εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά μα του 2017 είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια νέα πρόταση για ένα πιο ασφαλή μορφότυπο του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να λοιπόν, την έχουμε μπροστά μας την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεωρώ ότι βελτιώνει τα πράγματα, ενισχύει τις προδιαγραφές ασφαλείας του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου και επίσης συμβάλλει στην μείωση της πιθανότητας απάτης ή σε σχέση με το έγγραφο αυτό. Υπάρχει μια προθεσμία 15 Νοεμβρίου, με συγχωρείτε, για την κατάθεση αυτών των τροπολογιών. Η κυρία Κινίτσι και ο κύριος Δεπρέης και οι εισηγητές συμφώνησαν και αυτοί ότι δεν θα έπρεπε να υποβληθούν τροπολογίε και ότι θα έπρεπε να εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατό την πρόταση αυτή προκειμένου να κινηθούν γρήγορα και τα κράτη-μέλη και να εγκρίνουν και αυτά αυτή την πρόταση. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι προ το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Να καταφέρουν δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ταξιδιωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πρεσβείες και προξενία άλλων κρατών μελών. Εν τέλει, δεν καταφέραμε να αποφύγουμε τις τροπολογίες. Έχουμε 15 τροπολογίες. Εγώ δεν πρόκειται να εκπονήσω αυτή τη στιγμή συμβαστικές τροπολογίες. Θα τις θέσουμε τις 15 αυτές τροπολογίες προς ψήφιση. Θα δω και θα συζητήσω και με τους πιο ηγητές τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις τροπολογίες. Σε κάθε περίπτωση που παραλαμβάνω. Είναι πολύ σημαντικό να κινηθούμε γρήγορα, πολύ γρήγορα γιατί εδώ πέρα, αν θέλετε, έχουμε το, ένα καταπληκτικό παράδειγμα του πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στου πολίτε τη. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω του κοιόδη ε, εισηγητέ. Κίνγκα. Ε, σε ευχαριστούμε, Κίνγκα. Έχουμε την ψηφοφορία τον Δεκέμβριο και όπω είπατε, είναι ένα πολύ καλό πράγμα. τροπολογίε δεν ξέρω τι είναι. Θέλουμε κάποια περισσότερη αστριότητα εδώ, θέλουμε απλά να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω ημερομηνία. Κάποια στιγμή το Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ήθελε κάποιο άλλο να μιλήσει για τα επίγοντα ταξίδια. έγγραφα. Κάποια τροπολογία. Α, ναι. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ, Κλώτ. Ήθελα να παρέμβω κυρίως για το εξής, να ευχαριστήσω την κυρία Γκάλ και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την ε, δουλειά που έκαναν για να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα στο συντομότερο ε, διάστημα για το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι είχε αποφασιστεί άτυπα μεταξύ των σκιωδών εισηγητών να μην υποβάλουμε τροπολογίες για να πάμε πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, δύο συνάδελφοι υπέβαλαν τροπολογίες και προφανώς ε, και εγώ σεβόμενη την συνάδελφο Ε, θα μιλήσουμε βέβαια για τα ζητήματα αυτά, αλλά δεν θα υποβάλω τροπολογίε. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά βεβαίω υπάρχουν και οι άλλε τροπολογίε οι οποίε αφορούν την ε, καταστροφή του εγγράφου αυτού για λόγους οι οποίοι αφορούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης της ισχύω των εγγράφων αυτών σε περιπτώσεις επαναπατρισμού και ειδικά από ζώνες του κόσμου όπου υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε περαιτέρω το πεδίο της συζήτησης που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και είμαι σίγουρη ότι σε ένα πνεύμα συνεργασίας θα διευκολυνθεί η έγκριση αυτού του εγγράφου και θα αναζητήσουμε την καλύτερη λύση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όπως είπα λοιπόν θα συνεργαστούμε σε αυτό το πνεύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα, συγγνώμη, πρέπει να πω ότι είσαι σκιώδηση των των Σοσιαλδημοκρατών. Ε, Βεβαίω, εργαστήκε και εσύ σκληρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα, Κίνγκα. Αυτά. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Όχι, ωραία. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Πάει αυτό το θέμα. Περνάμε τώρα στο σημείο 8, εμπορία και χρήση πρόδρομων ε, εκρηκτικών. Θα ακούσουμε τον κύριο Μάμικινς, ο οποίος ε, θα μας παρουσιάσει τις 95 τροπολογίες, οι οποίες στηρίζουν ε, κυρίως την έκθεσή σας. Οπότε, Αντρέη, έλετε να μας πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Ε, η προθεσμία ήταν στις 5 Νοεμβρίου, είχαμε λάβει μέχρι τότε 72 τροπολογίες. Μετά την εξέταση των τροπολογιών μπορώ να πω ότι κυρίως ε, οδηγούν σε μια σύγκληση που ενισχύει τον ρυθμιστικό αντίκτυπο της πρότασης. Οι προτάσεις αυτές επίσης αντικατοπτρίζουν τις κύριες ιδέες που εκφράστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 18 Οκτωβρίου. Οι τροπολογίες ήδη έχουν περάσει από την ε, διαδικασία εξέτασης από την ε, νομική υπηρεσία και βρίσκονται προς μετάφραση. Αναμένω η μετάφραση να είναι έτοιμη για τις 23 Νοεμβρίου. Κάτι το σημαντικό αφορά τους αγρότες ε, ε, ως επαγγελματίες χρήστες και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρίσμπεκ που το πρότεινε καθώς έτσι υπάρχει σαφήνεια στον ορισμό. Επίσης αυτό ανταποκρίνεται και στην θέση του Συμβουλίου και επιπλέον η κυρία Γκρίσμπεκ συνεισέφερε και στον ορισμό των ύποπτων συναλλαγών που επίσης θεωρώ ότι είναι πολύτιμος. Όμως θα επιμείνω στην 24ωρη υποχρέωση αναφοράς ε, ύποπτων συναλλαγών, εάν θέλουμε να έχει κάποιο νόημα αυτή η διάταξη, πρέπει ε, η προθεσμία να είναι 24 ώρες. Και, και αυτό πολύ είναι. Όπως ξέρουμε, ο χρόνος ε, παίζει μεγάλη σημασία, χρειάζεται μισή ώρα ένας έμπειρος άνθρωπος να δημιουργήσει μια βόμβα από τα υλικά αυτά. Επίση, εκεί όπου βλέπω μια λογική συμφωνία, είναι η συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών φορέων σε όλες τις αγορές στο διαδίκτυο όσον αφορά τις υποχρεώσεις αναφοράς. Αυτό μας επιτρέπει να προστατεύσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την σχετική αγορά από τις σκιώδεις διαδικτυακές αγορές. Επιπλέον, κάποιοι βουλευτές είχαν υποβάλει σημαντικές προτάσεις της Κομισιόν για να υιοθετηθούν κατευθυντήριες γραμμές, κάτι το οποίο βρίσκω θετικό. Κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να συστήσουμε αφορά το άρθρο 15 και συγκεκριμένα την άδεια της ε, Κομισιόν ε, να εγκρίνει με πράξεις ε, κάτι εξουσιοδότηση αλλαγές στο παράρτημα ένα που αφορά τις ουσίες καθώς στόχος του κανονισμού είναι ακριβώς να μπορούμε να αντιδράσουμε καλύτερα στις νέες συνθήκες. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τι είναι η δυνατότητα της εποπτείας των πράξεων εξουσιοδότηση. Οπότε εδώ πέρα θα κερδίσουμε μόνο εάν κομισιόν, μπορούμε να παρεμβούμε, συγχωρείτε, μόνο εάν κομισιόν προσθέτει νέες ουσίες ε, και αυτό μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα. Και πολλές τροπολογίες είναι σχεδόν ταυτόσιμες. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι η ζωή μας θα γίνει πολύ πιο εύκολη. Και επιπροσθέτως ε, να σας ενημερώσω ότι είχα μία συνάντηση με τον Επίτροπο Κίνγκ στην ε, συνάντησή μας στην συνεδρίαση της Δευτέρας Οκτωβρίου και η Κομισιόν είπε ότι έχει κρίσιμη σημασία να δούμε το θέμα του σκοτεινού δικτύου. όπου εκεί πέρα γίνεται το παράνομο εμπόριο εκρηκτικών και τονίζει την σημασία των πράξεων κάτω εξουσιοδότηση ως ένα σημαντικό μέσο ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα. Στήριξε το σχέδιο έκθεσης, όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα, όμως δεδομένου του ότι πλησιάζουμε στο τέλος ε, της νομοθετικής μας ε, θητείας, Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο σωστά. Γι' αυτό προτείνω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια τεχνική συνάντηση για να είναι έτοιμο το κείμενο να ψηφιστεί στις 10 Δεκεμβρίου όπως προγραμματίσαμε. Και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο και μετά ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Ε, για το Συμβούλιο η εντολή της Κορεπέρ ε, υπολογίζεται να δοθεί στις 12 ε, Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι κύριε Πρόεδρε. Σας δίνω ξανά τον λόγο για να παρέμβουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Αντρέης. Θα ήθελα να μιλήσεις και εκ μέρους του σκιωδούς εισηγητού του ΕΛΚΑ συνάδελφου ναι, ο κύριος και μου είπε ότι μπορώ να του διαβάσω ε, ε, τις θέσεις του, ότι πρώτα πρώτα είναι θετική και με το παραπάνω αυτή η πρόταση, γιατί έχουμε αυτή την αύξηση των κριτικών και υπάρχουν σε τεχνικές για βόμβες, οπότε θα πρέπει να έχουμε ε, επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την πρόσβαση σε αυτές τις ουσίες, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους ε, ελέγχους και θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός αναφορά στις αρχές για τις δραστηριότητε. Επίσης έχουμε συζητήσει με πληροφοριών μυστικές υπηρεσίες, στους ε, επαγγελματίες του κλάδου. Οπότε ο κ. Στεχόφσκι λέει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε αύξηση της γραφειοκρατίας σχετικά. Ε, πάντως ε, πάρα πολύ θετική πρόταση και ελπίζει ότι θα υπάρξει ευρεία συνένεση για αυτό το σημαντικό για την ασφαλεία μα θέμα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ναταλή, για την Άλντε. Είσαι ηγήτρια, θες το λόγο. Κλώτης, ευχαριστώ. Δύο λόγια όσον αφορά τις τροπολογίες για αυτό το τόσο τεχνικό θέμα. Ε, όπως είπαν οι συνάδελφοι, είναι τεχνικό αλλά πολύ σημαντικό. Είναι θέμα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, πρόληψης των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων. Ε, ξεκινούμε από το θέμα ε, της ρεστιχνικής κατασκευής βομβών και όπως ελέγχθη θέλουμε ταυτόχρονα να πετύχουμε δύο στόχους να υπάρξει ένα ξεκάθαρος ορισμός και ανταλλαγή πληροφοριών των εμπλεκομένων δηλαδή της βιομηχανίας επίσης όλοι όσοι θα εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό. Θα πρέπει να υπάρχει γνώση της νομοθεσίας ε, και θα πρέπει να είναι εύκολη η εφαρμογή του κανονισμού. Μας είπε ο εισηγητής τα θέματα του ορισμού της ύποπτης συναλλαγής. Ε, θα είναι αυτό σημαντικό γιατί τότε θα συντρέχει η εφαρμογή του νομοθετήματος και των παραρτημάτων. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί μια συγκεκριμένη κατηγορία τέτοιων εκρηκτικών για τους γεωργούς. Αυτό θα το επεξεργαστούμε πριν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή. Επίσης, όσον αφορά τις ε, ανταλλαγές, στις τροπολογίες, προσπάθησα να προσθέσω την ιδέα των τακτών ε, ανταλλαγών μεταξύ των κατασταλτικών αρχών, των ελεγκτικών αρχών, των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων της ε, αγοράς και στο ίντερνετ, ε, πάντα επαγγελματία που εμπλέκεται για να υπάρξει αγαστή συνεργασία, κατανόηση και ορθή εφαρμογή του νόμου. Τώρα όσον αφορά τα εθνικά σημεία επαφής, πολύ σημαντικό να έχουμε μια πλατφόρμα ενημέρωσης ε, των οικονομικών φορέων, όλων που καλύπτουν τον κανονισμό. Με τις τροπολογίες επίσης προσπάθησα να ξεκαθαρίσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία ως κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή το πώς θα μπορούμε καλύτερα να αναγνωρίσουμε και να ε, ε, επισημαίνουμε αυτές τις υποτές συναλλαγές για αυτές τις πρόδρομες ουσίες των εκρηκτικών. Πώς θα περιβάλλει το λοιπόν, με περισσότερη ασφάλεια άπαξ η ουσία έχει αγοραστεί. Επίσης για τις τροπολογίες έχουμε εδώ ένα κανονισμό. Επομένω θα υπάρχει άμεση εφαρμογή στο ιστορικό των χωρών μελών. Είμαστε συνομοθέτες, άρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα το κείμενο, να έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα το είπε. Ναι, και εγώ να καταργηθεί η προθεσμία των 24 ωρών και να έχουμε ανταυτού το ταχύτερο δυνατόν ως διατύπωση. Να το συζητήσουμε βέβαια. Δεν αρκεί να μας αρέσει το κείμενο, αλλά θα πρέπει να είναι και εφαρμόσιμο από τους εμπλεκόμενους όσον αφορά την πώληση τέτοιων ουσιών που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες όταν χρησιμοποιηθεί και επίσης συμφωνώ με τα βασικά στοιχεία της πρώτας όπως είπε ο συγητής μας ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση αυτών που αγοράζουν τις πρόδρομες ουσίες ότι από τον κανονισμό ότι ορίζουν τα παραρτήματα Έχουμε και τη συνεργασία βέβαια με τον κύριο Κίνγκ για την προβληματική του σκοτεινού ίντερνετ, της αγοραπολισίες πιόνται εκεί, οπότε μπαίνει πάλι θέμα ε, επισήμανσης και εντοπισμού των υπόπτων ε, συναλλαγών. Καλά, αφού δεν με περιορίζετε, συνεχίζω. Ελπίζω να συνεχιστεί η αποτελεσματική μα και θετική συνεργασία και έτσι να καταφέρουμε ψήσουμε το κείμενο Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Ανταλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο πάλι έχει ο εισηγητής. Μάλλον, συγγνώμη, Μπόντιλ. Μπόντιλ Μπολέρο, θέλει το λόγο. Είσαι και εσύ όδη εισηγήτρια για τους πράσινους. Έχεις το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ απλά παίρνω το λόγο για να πω ότι η πολιτική μου ομάδα είναι υπέρ τη πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώ θα πρέπει να ενισχύσουμε την νομοθεσία για τι πρόδρομε ουσίε εκρηκτικών υλών, για να καταφέρουμε να αποφύγουμε τι τρομοκρατικέ επιθέσει, αλλά για να αποφύγουμε και κάτι ακόμα, την μόλυνση, την ρήπανση που προέρχεται από τι χημικέ αυτέ ουσίε. Έχουμε καταθέσει μια σειρά τροπολογιών που έχουν ως στόχο να αποσαφηνίσουν περισσότερο αυτό το οποίο ονομάζουμε επιγραμμική αγορά αγορά δηλαδή στο διαδίκτυο, μια ενδιάμεση αγορά διαδικτυακή και επίσης μέσω των τροπολογιών λέμε ότι θα πρέπει να συλλέγουμε περισσότερα δεδομένα για κάθε καταναλωτή που αγοράζει τέτοιες ουσίες. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε βέβαια αυτό να το επιτύχουμε στην πράξη. Προβλέπεται αυτή τη στιγμή ότι θα συλλέγονται και θα διατηρούνται τα δεδομένα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μαζικά όμως δεδομένα. Αυτό για μας προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, λέει ο κύριο Τερικάμπρα. Δεν άκουσα τη διερμηνία. Μήπω θέλει να το πω και στα αγγλικά, λέει η κυρία Μποντίλα. Δεν λειτουργήσε η διερμηνία, λέει ο κύριο Τερικάμπρα. Είχα συνδεθεί με την αγγλική διερμηνία, με το αγγλικό κανάλι και δεν μπόρεσα να ακούσω τη διερμηνία. Κύριε Ριγκάπρα, θέλει να ξανακούσετε την παρέμβαση. Η κυρία Μποντήλ είπε βασικά ότι δεν είμαστε κατά τη πρόταση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω τη πρόταση αυτή να αποφύγουμε μελλοντικέ τρομοκρατικέ επιθέσει, αλλά και να προστατεύσουμε το περιβάλλον λόγω τη ρήπανση που προκύπτει από τη χρήση των χημικών αυτών ουσιών. Λέω επίση ότι για ένα χρόνο θα πρέπει, θα πρέπει να ξαναδούμε το αν για ένα χρόνο πρέπει να διατηρούμε τις πληροφορίες αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες αυτές και τίθεται ένα ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πολύ ωραία, λειτουργεί η διερμηνία, λέει ο πρόεδρος. Άντρε, ο εισηγητής, θέλεις να πάρεις το λόγο, να καταλήξει κάποια συμπεράσματα. Δεν θέλω να πω σπουδαία πράγματα, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω απλώ τους και όδης για την πολύ καλή συνεργασία και συνεχίσουμε στον δρόμο αυτόν. Ωραία, σε ευχαριστούμε και εμείς πολύ. 10 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Προστασία του προπολογισμού τη Ένωση σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτο δικαίου στα κράτη-μέλη. Ανταλλαγή απόψεων για τι τροπολογίε. Συντάκτη γνωμοδότηση είναι ο κύριο Κάμπρα. Έχουμε εδώ πέρα μια πρόταση κανονισμού. Η ΛΥΜΠΕ, η επιτροπή μα, είναι συνδεδεμένη επιτροπή. Η Επιτροπή μας, αγαπητοί συνάδελφοι, δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα αυτό, καθότι είχαμε πολλές προκλήσεις και εξελίξεις όσον αφορά το κράτος δικαίου πρόσφατα και τίθεται το ζήτημα της προστασίας και της προώθησης των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λόγο τώρα έχει ο συγητής για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του και να μας παρουσιάσει κυρίως τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για τη γνωμοδότηση αυτή. Κύριε Τερικάμπρας, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Την προηγούμενη Τετάρτη, κύριε Πρόεδρε, έφτασε η τελευταία τροπολογία για τη γνωμοδότηση αυτή και συνολικά έχουμε 144 τροπολογίες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είχαμε τον απαραίτητο χρόνο να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Αξιολογήσαμε και κοιτάξαμε γρήγορα τις κατατηθήσεις τροπολογίες και έγινε μάλιστα και μία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών κατά τη διάρκεια της οποίας οι συνάδελφοί μου εξέφρασαν ανησυχίες, είπανε με ποιε τροπολογίε συμφωνούν και εν γέννη θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο όλοι μας και ότι θα καταφέρουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα τελικό πολύ καλό κείμενο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πρόταση που έχει εγκριθεί από όλου και μια άλλη πρόταση που είναι πιο αμφιλεγόμενη. Το πιο αμφιλεγόμενο, αν θέλετε, σημείο είναι αυτό που έχει να κάνει με την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, του προτινούμενου αυτού κανονισμού. Δηλαδή, να μην αφαιρόμαστε μόνο στο κράτος δικαίου, αλλά και στη δημοκρατία και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Μόλον ότι γνωρίζουμε ότι από νομικής πλευράς υπάρχει δυνατότητα αυτή εγώ αυτό, λέω, αυτό το οποίο λέω είναι ότι ε, το πιο σημαντικό είναι να εργαστούμε μέσω του, νομι... του κράτους δικαίου και μέσω του κράτους δικαίου ασχολούμεθα και με τη δημοκρατία και με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορεί λοιπόν το πεδίο εφαρμογή να είναι ευρύτερο και πάλι μπορούμε να επιμένουμε και με ένα πιο ευρύτερο πεδίο εφαρμογή σε αυτό που μα ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή στο κράτο δικαίου. Αλλά είναι ακόμα αμφιλεγόμενο το σημείο αυτό δεν συμφωνούν όλοι και οι θα πρέπει να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. Τώρα, το δεύτερο σημείο που το οποίο όλοι συμφωνούν είναι η δημιουργία ενός πάνελ εμπειρογνωμόνων. Υπάρχει μια σημαντική ανησυχία. Το ότι οι τελικοί δικαιούχοι, αν θέλετε, του κοινοτικού προπολογισμού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν ε, τα θύματα μιας κακής διαχείρισης διοικητικής εξαιτία ενός κράτους μέλους. Δεν θα πρέπει δικαιούχοι των προγραμμάτων να καταβάλουν το τίμημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό για να προστατεύσουμε τους δικαιούχους αυτούς, για να προστατεύσουμε τους ευρωπαίους πολίτες. Προκειμένου όμως να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ουδέτερο πάνελ εμπειρογνωμόνων Προφανώ θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μόνο τη σύνθεση λίγο του πάνελ αυτού, ποιοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο πάνελ αυτό, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει το πάνελ αυτό εμπειρογνωμόνων, ένα ουδέτερο πάνελ, αυτό θα αποτελέσει πολύ θετικό βήμα και κατά πάσα πιθανότητα θα διασκεδάσει οποιαδήποτε ιδεολογική, πολιτική, υπόνοια, επιρροής μπορεί να υπάρχει στη λήψη δύσκολων αποφάσεων. Επ' αυτού πάντως συμφωνούμε όλοι και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον, γιατί θα πρέπει να καταλήξουμε και σε μια σειρά συμβαστικών προτάσεων, προκειμένου να προωθήσουμε την πρόταση αυτή ακόμα περισσότερο. Πάντως είμαι πεπισμένος ότι θα τα καταφέρουμε και πραγματικά οι σκιώδεις εισηγητέ είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, φιλικοί, πολύ καλοί και ευφιέστατοι. Είμαι πεπισμένος λοιπόν θα καταλήξουμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. But the nice people you were talking about the shadows. Was it οι καλοί άνθρωποι για τους οποίους μιλάτε είναι και Μάλιστα. Ωραία. Ποιος από αυτούς τους καλούς ανθρώπους θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Αντάμοφ για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρόεδρε. Αντέμοφ. εκπρόσωπο τον κύριο Ράντεφ, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής. Ε, δυστυχώς η πτήση του καθυστέρησε. Συμφωνούμε όλοι ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προστατευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γι' αυτό έχουμε τη διαδικασία του άρθρου 7 των συνθήκων Το σχέδιο έκθεσης και οι τροπολογίες που συζητάμε σήμερα προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό που δεν έχει νομική βάση. Αντί να αναφέρουμε ε, μια ξεκάθαρη θέση και σχέση μεταξύ αυτών των ζητημάτων, να ασχολούμαστε με ζητήματα που δεν έχουν νομική βάση. Γι' αυτό ζητάω από τους ε, συναδέλφους ε, να ξανασκεφτούν εάν θέλουν ε, να στηρίξουν μια έκθεση η οποία θα απορριφθεί ως παράνομη ή να ευθύσουν μια απόφαση η οποία δεν θα οδηγήσει σε απώλεια χρηματοδότησης για τους τελικούς δικαιούχους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και ο Γιούρεκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ε, είμαι σίγουρος ε, για το εάν θα βοηθήσει η καλή ατμόσφαιρα να σπάσει ο παγός, ε, γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως ε, όταν έχουμε τόσο συμπαθείς συναδέλφους ε, μπορούμε να ξεπεράσουμε ευκολότερα τις διαφορές. Διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν ε, σοβαρές αμφιβολίες. Δείτε τον τίτλο του ψηφίσματος. γενικευμένες ελλείψεις λέει εδώ πέρα, πολύ γενικόλογο. Δεν αφορά κάτι το συγκεκριμένο το οποίο αφορά την λειτουργία του κράτους ε, δικαίου γιατί βεβαίως ε, τα κανονικά ας πούμε, προβλήματα είναι αντικείμενο του δικαστηρίου. Αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε πρόταθεί οι αποφάσει του δικαστηρίου να επηρεάζουν τον προπολογισμό. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα ερώτημα. Με ποιον κανόνα μπορούμε να πούμε ότι στην χώρα Α υπάρχουν γενικευμένα προβλήματα κράτους δικαίου όταν η συνθήκη στο δεύτερο άρθρο λέει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής είναι δημοκρατικές χώρες και το να αρνηθούμε κάτι τέτοιο γίνεται μόνο με βάση την διαδικασία του άρθρου 7. Αν έχουμε άρθρο 7 είναι σαφές. Τα συμβαλόμενα μέρη θα πούν ότι μία από τις χώρες ε, παραβίασε αυτούς τους κανόνες, αλλιώς κάθε ένας έχει την απόψή του. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πει ότι δεν αποτελείται από δημοκρατικές χώρες, ε, τότε ερμηνεύουμε τα πράγματα κατά το δοκούν. Και μετά τα πράγματα είναι στα χέρια των κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τρεις αρχές ε, που μπορούν να πούν ότι έχει παραβιαστεί το άρθρο 2. Δηλαδή το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, με συγχωρείτε, Κομισιόν ή το 1 τρίτο των κρατών μελών. Ας φανταστούμε δηλαδή ότι κάποιο κράτος μέλος ε, ε, κάνει κάτι τέτοιο. Οι 10 χώρες λοιπόν αυτές δεν έχουν προπολογισμό. Τι θα κάνουν. Θα περιορίσουν το ελεύθερο εμπόριο, την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Μπαίνουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια μετά. Και κάτι άλλο. τονίζει την ειλικρίνεια του ε, εγχειρήματο αυτού. Ο καθηγητής Τερακάμπρα είπε ότι πρέπει να το διαμορφώσουμε έτσι ώστε να μην υποστούν οι πολίτες τις συνέπειες. Ε, αυτό λοιπόν διαψεύδει αυτό το οποίο ακούμε συχνά. Γιατί μας λέτε ότι η επίθεση σε ένα κράτος δεν είναι επίθεση στους πολίτες του. Ε, δυστυχώς, η επίθεση σε μια κυβέρνηση που εξέλεξαν οι πολίτες θα βλάψει τους πολίτες. Πρέπει να σκεφτούμε τα επιχειρήματα και να εξετάσουμε τις απόψεις. Θα σκεφτούμε πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι στο κράτος μέλος Α έχει παραβιαστεί η δημοκρατία. χωρίς απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια βάση. Ευχαριστώ. Η Σόφη για την Άλτε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη παρέμβαση νομίζω τονίζει γιατί χρειαζόμαστε έναν τέτοιο μηχανισμό. Ο κύριος Γιούρεκ και εγώ διαφωνούμε, αυτό είναι γνωστό. Εγώ δεν θεωρώ ότι η δημοκρατία είναι απλά η άποψη της ε, πλειοψηφίας ε, ή της κοινοβουλευτικής ε, πλειοψηφίας, δεν είναι αυτό η δημοκρατία. Και δεν είναι οπωσδήποτε το κράτος δικαίου. Είναι μια δικτατορία της πλειοψηφίας. Δεύτερον, εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση ισούται με τον λαό. Όλα όμω είναι κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση και κατά την άποψή σα, αυτή τη στιγμή κάποιο έχει καταλάβει την εξουσία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι βλέπετε εσείς την δημοκρατία και νομίζω ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουν να αντιλαμβάνονται γιατί χρειαζόμαστε μηχανισμό για να διασφαλίσουμε το δημοκρατικό κράτος και τα θεμελιώδη δικαιώματα εντό της Ένωσης. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό, καταλαβαίνω ότι αυτό βεβαίως ε, ενοχλεί κάποιες κυβερνήσεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Τώρα για το μέσο αυτό της αιρεσιμότητας ε, έχω κάποια ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας πολύ ρεαλιστικός τρόπος να, κυβερνήσουμε τις κυβερνή... να τιμωρήσουμε τις κυβερνήσεις και να φροντίσουμε να τηρούν όλε τι ίδιες προδιαγραφές. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση υπογραμμίζει τους κινδύνους πρώτα απ' όλα μπλέκουμε συνεχώς την αιρεσιμότητα με τις κυρώσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και όμως μιλάμε για την αιρεσιμότητα σαν να μιλάμε για κυρώσεις. Δεύτερον, Βεβαίω, αν και είναι απολύτως φυσιολογικό να περιμένουμε τα κράτη-μέλη που δέχονται χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχονται όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 2, οπότε σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ. Αλλά εάν είναι να χρησιμοποιηθεί για κυρώσεις ή πίεση στα κράτη-μέλη, τότε κινδυνεύει να είναι άδικο. Γιατί βεβαίως ε, γνωρίζουμε ότι οι καθαροί εισφορείς δεν θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τις χώρες οι οποίες ε, λαμβάνουν ε, στον ισολογισμό χρήματα από την Ένωση και γνωρίζουμε ότι θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Τρίτον, απογοητεύομαι από το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει αυτή την πρόταση για να ξεφύγει από τον μηχανισμό τον σωστό που είχαμε προτείνει την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε ένα ψήφισμα. Ρυθμίζαμε την νομοθετική πρωτοβουλία και το περίεργο εδώ με την Κομισιόν είναι ότι όποτε το Συμβούλιο λέει θέλουμε κάτι γελίο, για το οποίο δεν υπάρχει νομική βάση ούτε κατά διάνοια, η Κομισιόν υποβάλλει μια πρόταση σε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΕΡΕΤΟ, ε, υποβάλλει μια έκθεση νοθική πρωτοβουλία, ε, η Κομισιόν την αγνοεί. Οπότε, αντί να υποβάλει έναν κανονικό μηχανισμό όπου η ιδιοκτησία των αξιών της Ένωσης θα είναι στα χέρια των πολιτών και των εκπροσώπων του στα Εθνικά Κοινοβούλια και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση η οποία ουσιαστικά δίνει την εξουσία σε κάποιους δημοσίους υπαλλήλους. Ε, Μου αρέσει αυτή η φράση, αλλά εδώ πέρα αυτό ισχύει. Θα τσεκάρει κάποιος ένα κατάλογο ένα ε, υπάλληλο αν είναι δυνατόν. Αυτό αντιβαίνει ε, όλα όσα πιστεύουμε. Οπότε και τα συναισθήματα. Καλωσορίζω το ότι ο εισηγητή αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή σε όλα αυτά, δηλαδή δημοκρατία, κράτο δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα που καλύπτει το άρθρο 2. Είναι αλληλένδετα. ζητήσατε να υπάρξει ένα πάνελ ειδικών. Παραδείγματος χάρη πηγαίνει στην κατεύθυνση αυτού που θέλει η Κομισιόν. Κάτι το τεχνοκρατικό, γραφειοκρατικό. Εγώ προτείνω, αν δεχτούμε αυτή την αιρεσιμότητα, πρέπει να διαμορφώσουμε τους όρους. Όχι να το κάνει η Κομισιόν όμως, πρέπει να υπάρχει μια δημόσια συζήτηση. Όπως είχαμε προτείνει εμείς το σχετικό πακέτο και προτείνατε ακριβώ να μπουν αυτές τι τροπολογίε στην συμβαστική σα πρόταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Okay. Right, Mr. Κύριε Γιούρεκ, θέλετε να επιχειρηματολογήσετε εναντίον. Ναι, ναι, ναι, πρέπει, πρέπει να αντιδράσω, γιατί μπορεί να φταίει η μετάφραση, λέει ο κύριος γιατί δεν νομίζω ότι ε, ήθελε να πει αυτά που άκουσα από τη μετάφραση η Σοφή ή ότι άκουσε όσα είπα εγώ σωστά, γιατί δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση ε, εγώ δεν ήθελα να ταυτίσω την κυβέρνηση με τους ε, πολίτες. Είπα μόνο ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία η κυβέρνηση εκπροσωπεί, εκπροσωπεί την πλειοψηφία των πολιτών. Και σε μια πλουραλιστική κοινωνία ε, είναι θεμητό να υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Οπότε θα πρέπει να ισχύουν και να ακούνται τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών. Και νομίζω ότι υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση στα όσα είπε η Σοφία γιατί συνεχώς εμένουμε στο ότι το Κοινοβούλιο η πλειοψηφία δεν σημαίνει ότι είναι αλάνθαστη γιατί άλλο πλειοψηφία, άλλο ειδική πλειοψηφία η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε την πλειοψηφία των χωρών ούτε την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό πιστεύω ότι ισχύει όσον αφορά τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος. Κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, λέει η κυρία Νιτφέλτ. Πρώτα-πρώτα. Όχι, η κυβέρνηση που έχει πλησιάσει στο Κοινοβουλίο δεν σημαίνει την πλειοψηφία των ψήφων του λαού. Το γνωρίζουμε αυτό. Και από την άλλη μεριά, πλειοψηφία δεν σημαίνει να κάνει κανεί ό,τι θέλει. Ο Πρόεδρο, α κλείσουμε το, την αντιπαράθεση. Μπορεί να λάβει το λόγο η κυρία Κέγκη, αν και ήρθε λίγο αργά, είναι εισηγητρία για το S&D, για τους σοσιαλδημοκράτες. Κλοντ, σε ευχαριστώ. Θα είμαι πραγματικά σύντομη και ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο νομοδοτήσεις και για τις ε, προσπάθειες που έκανε να πάσχει σε ένα συμβασμό στις πολιτικές ομάδες. Είμαστε κοινότητα δικαίου και οι αξίες μας είναι η βάση, το θεμέλιο της ύπαρξης. Και άρα η τήρηση αυτών των αρχών θα πρέπει να περιβάλλεται από εγγύσεις μέσω οποιασδήποτε πολιτικής και μέσω του προϋπολογισμού. Πολύ καλά τα δούλεψε, τα επεξεργάστηκε όλα αυτά ο συγητής όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής ε, και για την υποκατάσταση του κράτους δικαίου με τις αξίες της Ένωσης που έβαλε. Προς τα εκεί Και ο πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών κατεβάσαμε κάποιες τροπολογίες και εμείς με τη σειρά μας λέμε ότι το κράτος δικαίου σχετίζεται με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Αυτές είναι τρεις αξίες που είναι σαν ένα τρίγωνο. Ε, αλληλοσυνδέονται, δεν μπορεί να σταθεί μία αξία χωρίς άλλες δύο και είναι και το θέμα της νομικής βάσης οπότε και ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει ε, στο θέμα που κολλήσαμε η νομική μας υπηρεσία με έναν, ε, ε, με έναν μηχανισμό που να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό οπότε έχουμε καταπάτηση αυτών των αργών. και ελπίζουμε ότι όλοι μαζί θα μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβαστικό κείμενο. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε Σεσίλ, λέει ο Πρόεδρος. 3 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε εισηγητά για να κλείστε. και Τελικάμπρας. Πώς λέτε Πρόεδρε, υπάρχουν ζητήματα επίμαχα. Είμαι βέβαιος ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρόκειται να τα συζητήσουμε. Πολύ ωραία. Καλά που τα είπες έτσι συμβαστικά. Πρέπει να βιαστούμε γιατί έχουμε πολλά θέματα στη μέση διάταξη. Πάμε στο 20, λέει ο Πρόεδρος. Προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ευρωεκλογών. Πρόκειται για την ε, πρόταση οδηγία για την προστασία των δεδομένων, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, στη συνέχεια του σκανδάλου που ξέσπασε σε σχέση με το Facebook και την υπηρεσία και την εταιρεία και με τις αναλύτικα θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε όπως προβλέπει η διάταξη 53 και η συγκεκριμένη η έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση, δεν είναι εκτενές το κείμενο. Αναφέρεται πάντως σε ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά το σκάνδαλο Facebook Cambridge Analytica. Η πρόταση αυτή καταδεικνύει πλέον την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβει δράση. Αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας μηχανισμός, ένα μέσο επιβολής χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε πολιτικά κόμματα ή ιδρύματα, τα οποία σκεμμένα επηρεάζουν ή αποπειρώνται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Με εδώ ξεκινά για μένα το πρόβλημα όμως. Απόπειρα επιρροής εκλογών ή αποτελέσματος εκλογών, αυτό δεν λέγεται εκστρατεία. <laughs> Αυτό δεν κάνουμε όλοι μας. Επομένως το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τελικά ποιες δράσεις στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της. Δεν είναι σαφές αυτό για μένα. Και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια διαδικασία που ξεκινά με απόφαση μια υπηρεσία, προστασίας δεδομένων από την οποία φαίνεται ότι έχει γίνει μια παράβαση σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από πολιτικό κόμμα, από πολιτικό ίδρυμα και το Και περιγράφεται εν συνεχεία στο κείμενο η όλη διαδικασία. Έχω καταθέσει κύριε Πρόεδρε κάποιε τροπολογίε προκειμένου η προβλεπόμενη διαδικασία να είναι πιο συμπαγής από νομικής πλευράς. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα όσα προτείνονται δεν επιλύουν σε καμία περίπτωση το κεντρικό πρόβλημα το οποίο σας εξήγησα. Δηλαδή, δεν είμαι καθόλου σίγουρη τι θέλει να επιλύσει εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν ένα πολιτικό κόμμα έχει παραβιάσει τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, τότε τον κανονισμό αυτόν έχει παραβιάσει και θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις αν έχει παραβιάσει τους κανόνες που ισχύουν για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, προβλέπονται σχετικές διαδικασίες και εκεί. Επομένως, δεν είμαι πεπισμένη αυτή τη στιγμή για το ποιε δράσει θέλει να καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίε υποτίθεται ότι δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νοσιακή νομοθεσία. Αυτό είναι ένα εκρεμέ ερώτημα ακόμα για μένα. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Ενδεχομένω να φταίει το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει αξιολόγηση αντικτύπου. Μήπω θα έπρεπε να το κάνει αυτό και ουσιαστικά να δει ποιε τελικά εκθέσεις της δικής μας Επιτροπής συνοδεύονται από εκτίμηση αντικτύπου, γιατί νομίζω ότι ο αριθμός θα είναι μηδέν. Νομίζω ότι είμαστε από τις επιτροπές εκείνες του Κοινοβουλίου που αξιολογούν εκθέσεις προτάσει νομοθεσία, χωρί να έχει γίνει όμω καμία εκτίμηση αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, α προσπαθήσουμε λίγο να δούμε τι θέλουμε να επιλύσουμε με την προτινόμενη αυτή νομοθεσία. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι πρέπει να νομοθετούμε για τα σημαντικά μονοζητήματα και ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την περιττή νομοθεσία. Ας μου απαντήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επανέρχομαι στο αρχικό ζήτημα το οποίο έθιξα, ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εκκίνησης της προβλεπόμενης αυτής διαδικασίας και να μην κινείται η όλη διαδικασία όταν υπάρχει μόνο μία απόφαση από μία εποπτική αρχή για τα προσωπικά, προσωπικά δεδομένα. Τέλο πάντων, ακόμα και αν οι τροπολογίε μου καταστήσουν όλη τη διαδικασία λίγο πιο συγκεκριμένη και σαφή, παρόλα αυτά περιμένω απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ ωραία, Σόφη, σε ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε, γιατί ε, η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή ΑΦΚΟ και ο εκεί εισηγητή, η συγγήτρια μάλλον, φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί με τα πιο θεμελιώδη ζητήματα. Δηλαδή, ε, ποιο προβαίνει στην ε, πολιτική εκστρατεία, ποιο δημοσιεύει τι συγκεκριμένε διαφημίσει κτλ. Αυτό το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι όταν γίνεται μία απόπειρα επιρροής, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση του Facebook και της Cambridge Analytica. Αναφερόμαστε εδώ σε παράνομες δραστηριότητες. Δραστηριότητες οι οποίες θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ως παράνομες. Μπορεί να είναι νόμιμες σε μια δικαιοδοσία συγκεκριμένη. Ξέρετε ότι υπάρχουν κανόνες στις ΗΠΑ οι οποίοι δεν ισχύουν για την δικαιοδοσία, για την ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αντίστροφο. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, αποσπασματικά χρησιμοποιείται κάπως η νομοθεσία. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η ΑΦΚΟ είναι να δημιουργήσει ένα συμπαγές πλαίσιο όπου να γνωρίζουμε ακριβώς πλέον ποιοι είναι οι ηθήνοντες για τις ε, αθέμητες αυτές οι παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο των εκλογών. Νομίζω ότι η δική μα τώρα η Επιτροπή, ω πιο ειδικευμένη Επιτροπή, μπορεί να βάλει και αυτή το λιθαράκι τη, προφανώ για το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, αλλά και για πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξέρεις ότι ε, υπάρχει ένας κατάλογος δραστηριοτήτων που μπορεί να αντιστοιχεί σε μια προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται και μια σχετική αναφορά σε κάποιε τουλάχιστον από τι δραστηριότητε αυτέ. Επειδή εσύ είπε ότι όλα αυτά ουσιαστικά αποτελούν ε, προεκλογική εκστρατεία. Δεν είναι απλώ έτσι. Ναι, ναι, υπάρχει προεκλογική εκστρατεία και υπάρχει και η παράνομη δραστηριότητα. Αλλά αν κάτι είναι παράνομο, δεν χρειάζεται επιπλέον νομοθεσία. Αν κάτι είναι παράνομο, τότε γι' αυτό μπορούν να επιβληθούν κυρώσει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως παράνομες. Ακόμα και αν είμαστε υπεύθυνοι για ένα μικρό τμήμα τελικά της πρότασης, ας μην προχωρήσουμε ευσπεσμένα με την πρόταση αυτή μόνο και μόνο για να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε δραστήριοι. Μα δεν προχωράμε γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος, αλλά από την άλλη ζυγώνουν και οι ευρωπαϊκές εκλογές και από την άλλη είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι γίνονται απόπειρε επιρροή και των ευρωπαϊκών εκλογών. Απέναντι λοιπόν στο ζήτημα αυτό θα πρέπει κανείς να αντιδράσει γρήγορα αλλά και ποιοτικά. Μπορεί να μην σε έχω πείσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία επιφέρουν προς τη θέμενη αξία. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ, όπω είπα, θα ασχοληθεί κυρίως με το σκέλος εκείνο που έχει να κάνει με τις εκλογές και θα προσπαθήσει να δει η ΕΦΚΟ από πού πηγάζει η πολιτική διαφήμιση, η ε, εκλογική καμπάνια. Μολονότι εμεί ε, συντάσσουμε σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού μια σύντομη γνωμοδότηση, θεωρώ ότι η γνωμοδότησή μα θα είναι πολύ σημαντική. Ναι, αλλά αν μιλάς για στοχευμένη διαφήμιση, τότε δεν είναι λίγο περίεργο το ότι αναφερόμαστε τώρα στο ζήτημα αυτό, αλλά από την άλλη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θέλει να αναλάβει δράση για, την, για το e-privacy. Πρόσφατα νομίζω ότι κατέληξαν ενδεχομένω σε μια κοινή θέση, αλλά αν πραγματικά προχωρούσαν περισσότερο, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία έθιξε, Πρόεδρο. Ναι, αλλά ξέρει ότι ο κανονισμό GDPR δεν θα αντιμετωπίσει σκάνδαλα σαν αυτό του Facebook και του Cambridge Analytica. Είναι μέσω του e-privacy που θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια σκάνδαλα σαν αυτό τη Cambridge Analytica. Νομίζω λοιπόν ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν ε, να ενσωματωθούν στην γνωμοδότησή σου. Θα μπορούσες να κάνεις μία αναφορά στα ζητήματα αυτά στον περιορισμένο αριθμό λέξεων βέβαια που έχουμε εμείς για να γνωμοδοτήσουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ω Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να μπορούμε να αφαιρθούμε σε συγκεκριμένα μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Και βέβαια, όπω είπε και εσύ, η προτινόμενη νομοθεσία ή privacy θα αντιμετωπίσει μέρο τουλάχιστον των προβλημάτων που πηγάζουν από σκάνδαλα σαν αυτό του Facebook και τη Cambridge Analytica. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά θεωρώ ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι σημαντική γνωμοδότηση. Κύριο Σφόρτη, τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε. Να αντιδράσω απλώς αυτά που είπε η κυρία Σοφή Ιντβέλτ. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Μέσω του προτινόμενου αυτού μέσου, που έρχεται να συμπληρώσει ουσιαστικά την τροποποίηση που κάναμε φέτος στην υφιστάμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τους σωστούς κανόνες και τις σωστές κυρώσεις προκειμένου τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα να λειτουργούν νόμιμα, θεμητά, ισότιμα, χωρίς ε, να προβλέπονται περιπτώσεις ε, απάτης. Έχουμε κανόνες στα πλαίσια του GDPR στα πλαίσια του κανονισμού αυτού, οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα παραβιάζει τον κανονισμό αυτό, τον κανονισμό GDPR, θα το επιβάλλονται κυρώσεις. Ο στόχος όμως, η συγκεκριμένη αυτή πρόταση, έχει να κάνει περισσότερο με την περίπτωση πολιτικών κομμάτων ευρωπαϊκών που παραβιάζουν τον γενικό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου αθέμητα ή παράνομα να στοχεύσουν συγκεκριμένους ψηφοφόρους ή να προωθήσουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ξέρετε ότι ακόμα και αν έχουν παραβιάσει τον κανονισμό GDPR δεν πρόκειται να επομιστούν τα κόμματα αυτά κυρώσει που κανονικά θα έπρεπε να επιβληθούν από τον κανονισμό που υπάρχει για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων. Επομένω, δεν πρόκειται με άλλα λόγια να μειωθεί η χρηματοδότησή του. Εμεί θα θέλαμε να καταφέρουμε τώρα να στοχεύσουμε και τα κόμματα αυτά τα οποία παραβιάζοντα τον κανονισμό GDPR τελικά αθετούν, παραβιάζουν και τους κανόνες ε, για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και τελικά χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές στα πλαίσια μιας προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και το είπα έτσι γρήγορα, εν συντομία. Θα πρέπει όμως και εσείς τότε να διαβάσετε τη δική μα τη γνωμοδότηση, έτσι δεν είναι. Γιατί αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο είπε η συντάκτρια τη γνωμοδότηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κανονισμό GDPR από μόνο του δεν είναι τέλειο. Αυτό το οποίο όμως μας λέτε τώρα εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι στο πλαίσιο του GDPR δεν καλύπτονται επί του παρόντος τα εθνικά πολιτικά κόμματα και σχετική νομοθεσία, έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά τα πολιτικά κόμματα μπορούν να αναλάβουν δραστηριότητες μέσω του Facebook και μπορούν να προφήσουν κακόβουλο υλικό αν θέλετε το οποίο δεν καλύπτεται έπειτα από τον κανονισμό GDPR, έτσι δεν είναι αυτό, δεν μας είπατε. Σοφίντ Βέλτα, κοιτάξτε, δεν είμαι δικηγόρος, ιστορία σπούδασα, αλλά έμαθα να καταλαβαίνω δύο-τρία πράγματα περί νομικής ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλετε να επιβάλλετε κυρώσεις, θα πρέπει να ορίσετε με νομικούς όρους τι συνιστά παραβίαση. Θα πρέπει να ορίσετε με άλλα λόγια τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο κανονισμός GDPR δεν τηρήθηκε, παραβιάστηκε για, με κακόβουλο στόχο, με κακόβουλο σκοπό. Τι, τι εστί, τι σημαίνει κακόβουλο, αυτό θα πρέπει να το ορίσετε. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά πολιτικά κόμματα που χρησιμοποιούν τα κενά της νομοθεσίας για να κερδίσουν ολόκληρες εκλογές. Όλα αυτά με τρομάζουν πάρα πολύ, λέει η συγγήτρια. Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει ένα παράδειγμα. Μα κοιτάξτε, στα πλαίσια του κανονισμού GDPR ορίζονται και οι κυρώσεις και ορίζονται και οι παραβιάσεις οι περιπτώσει παραβίαση αυτού του κανονισμού. Αυτό το οποίο θέλουμε να στοχεύσουμε όμω με την πρόταση αυτή είναι ο τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παραβίαση του GDPR προκειμένου να επηρεάσουν με τρόπο αρνητικό την προεκλογική εκστρατεία για τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Δεν μπορεί να το κρίνει βέβαια αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθείται μια ολόκληρη διαδικασία την οποία την περιγράφουμε στην τροποποίηση αυτή της νομοθεσίας στα πλαίσια της οποίας τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να καθορίσουν, να αποφανθούν για το κατά πόσο έγινε παράνομη χρήση συγκεκριμένων πληροφοριών και στην περίπτωση αυτή θα επιβληθούν οι οι οποίες θα αναλογούν βέβαια με την χρηματοδότηση την οποία έχουν πολιτικά κόμματα. Δεν δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι δύο φορές θα επιβληθούν κυρώσεις σε ένα κόμμα για παράδειγμα. Θα επιβληθούν κυρώσει από το GDPR και θα επιβληθούν επιπλέον κυρώσει από τη νέα αυτή πρόταση. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό, δεν νομίζω ότι στέκει από νομικής πλευρά θα πρέπει πραγματικά να ορίσετε, όπως σας το είπα, ποια ήταν η κακόβουλη πρόθεση του συγκεκριμένου κόμματος. Με την εξαίρεση βέβαια του δικού μου πολιτικού κόμματος, <laughs> όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα είναι κακόβουλα, έτσι δεν είναι, εφόσον διαφωνώ με αυτά. Πολύ εύκολο λοιπόν να τα χαρακτηρίσω κακόβουλα. Είναι επικίνδυνο κάπως αυτό το οποίο προτείνεται, γιατί ε, ουσιαστικά προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να καθορίσετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μπορούν να κάνουν και τι όχι τα πολιτικά κόμματα, τι μπορούν να διατείνονται στη τελευταία ανάλυση, τι μπορούν να λένε προ τα, έξω και τι όχι. Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση θα φροντίσω να προσαρμόσω κατάλληλα τη γνωμοδότησή μου, λέει κυρία Εντβέλτ. Προχωρήσω παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ε, λυπάμαι που σας διακόπτω. Αλλά σας ευχαριστώ και καλή τύχη. και ευχαριστώ και την Κομισιόν. Ελπίζω να το συζητήσουμε και άλλο το ζήτημα. Τι μα είναι εφιάλτης αυτά τα πράγματα. Να τα συζητάμε σε δύο λεπτά. Τέλος τελείωσε τώρα. Περνάμε στο σημείο 11. επάρκεια της συμφωνίας με την Ιαπωνία. Ε, ο χρόνος ε, έχει τελειώσει. Τι κάνουμε, ακόμα κατευθύνει την Κομισιόν. Λοιπόν, συνάδελφοι, το επόμενο θέμα είναι η συμφωνία με την Ιαπωνία. Λοιπόν, η Κομισιόν έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο εφαρμοστική απόφαση για το επαρκέ επίπεδο προστασία που παρέχει η Ιαπωνία. Πρόκειται για την πρώτη σχετική απόφαση σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR. Οι συντονιστέ αποφάσισαν στι 27 Σεπτεμβρίου να προετοιμάσουν ένα σχέδιο ψηφίσματο για να εκφράσουν τι απόψει και τα σχόλια τη ΛΥΜΠΕ σε σχέση με το σχέδιο εφαρμοστική απόφαση που υπέβαλε η Κομισιόν. Το έγγραφο το προετοιμάσαμε έχοντας ε, λάβει υπόψη τις συνεισφορές των πολιτικών ομάδων και βεβαίως ε, λέει πως ε, είναι επαρκής η Ιαπωνία αλλά απαιτούνται κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά πολλά και σημαντικά ζητήματα ακριβώς για να δούμε τις διαφορές πτυχές του νομικού πλαισίου της Ιαπωνίας και να υπάρχει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας όπως απαιτεί το δικαστήριο. Λοιπόν, θα δώσουμε τον λόγο στα μέλη, ξεκινώντα από του κοιόδησηγητέ. Κύριε Κοέλιο, περιμένετε εκεί υπομονετικά, παρακαλώ λοιπόν. Ευχαριστώ. Είμαι και εγώ σκιοδησηγητής εξ ονόματος του κυρίου Μπόνη. Σας ευχαριστώ και αναμένουμε την περαιτέρω συνεργασία. Ο κύριος Μπόνη θέλει να τονίσει ότι η απόφαση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα. Και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τρίτη χώρα προχωρούν σε μια αμοιβαία αναγνώριση ισοδύναμου επίπεδου προστασίας και του άρθρου 45. Αυτό θα δημιουργήσει την μεγαλύτερη περιοχή ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων στον κόσμο και έτσι οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα από και προς την Ιαπωνία και ταυτόχρονα θα υπάρχει και πρόσβαση στην αγορά. Και βέβαια αναμένεται να ενισχύσει τις εμπορικέ και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν το σύστημα της άλλης επαρκές ε, και συμβατό. Έτσι θα επιτραπεί ασφαλής ροή δεδομένων μεταξύ των δύο πλευρών χωρίς ε, να υπάρχουν επιπρόσθετες διασφαλίσεις. Για να εγγυηθεί ένα ισοδύναμο επίπεδο, η Ιαπωνία συμφώνησε να υπάρξουν κάποιες επρόσθετες διασφαλίσεις. Προσφάτως εξυγχρόνισε τη σχετική της ε, νομοθεσία και την σύγκληση μεταξύ των δύο συστημάτων. Και βεβαίως ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ε, αυτό. Η Ιαπωνία άλλαξε το δικαιό της, αναγνωρίζει πλέον ε, την προστασία της ιδιωτικότητας ως εμελιώδες δικαίωμα. Και βεβαίως έχουμε εδώ πέρα παγκόσμια προδιαγραφή που ίσως υιοθετηθεί και από άλλες ε, χώρες για να έχουν ακριβώς ασφαλείς μεταφορές ε, δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπόνι θεωρεί ότι το σχέδιο ψηφίσματος ε, στην τρέχουσα μορφή του θα στείλει το λάθος μήνυμα και βεβαίω ε, θα πρέπει να υπάρχει και επαρκής προστασία με ισοδυναμούς κανόνες και είναι σαφές ότι από την ευρωπαϊκή πλευρά θέλουμε να διασφαλίσουμε σεβασμό του GDPR και ότι θα είναι μεταφορές, ε, δυνατές οι μεταφορές εκτός της Ευρωπαϊκής μόνο αν υπάρχει επαρκής προστασία. Βεβαίω, το θέμα αφορά την ισοδυναμία και όχι την απόλυτη ταύτιση. Οπότε θέλουμε ακριβώς να στείλουμε το μήνυμα του ότι εξετάζουμε την διαδικασία χωρίς να είμαστε υπερβολικά επικριτικοί, κάτι το οποίο θα φανεί και από τις τροπολογίες του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Σόφη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ σχεδόν με όλα ε, πάντα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερο επικριτικοί σε αυτό, διαφωνώ. Αλλά πολλές από τις ανησυχίες ε, που είχαμε καλύφθηκαν ε, το σχέδιο έκθεσής σας και βεβαίως θα εξετάσουμε με κριτική ματιά το θέμα αυτό και το τελικό κείμενο. αλλά νομίζω οι γενικέ γραμμές αντικατοπτρίζονται οι ανησυχίες μας. Θα δώσω τον λόγο στην Κομισιόν, αλλά πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε λάβει ήδη κάποια σχόλια από την νομική υπηρεσία ότι θα εξετάσουν το θέμα αυτό σε μια τεχνική συνάντηση. Θα το εξετάσουμε. Κύριε Τζεν Καρέλη, λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την τεχνική συνάντηση αυτή. Και πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για το ότι αντιλαμβάνεστε την σημασία των ευρημάτων αυτών. Δεν πρόκειται μόνο για την πρώτη συμφωνία επάρκειας του GDPR, αλλά και την πρώτη συμφωνία με χώρα που άλλαξε την προσέγγιση της και αποφάσισε να ακολουθήσει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλα τα βασικά της στοιχεία με ανεξάρτητη αρχή και τα λοιπά. Και πρώτη, για την πρώτη απόφαση ισοδυναμίας που αφορά μια μεγάλη χώρα της Ασίας και του Ειρηνικού που περιττώ να πούμε ότι είναι μια περιοχή του κόσμου με τεράστια στρατηγική σημασία αλλά βεβαίως ε, είναι και η πρώτη απόφαση που θα εφαρμόσει τη νέα προσέγγιση της Ένωσης για την ροή των δεδομένων που ζήτησε το Κοινοβούλιο, δηλαδή ότι δεν θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ότι θα πρέπει ακριβώς να χρησιμοποιηθούν τα μέσα GDPR για να υπάρξει ε, ελεύθερη ροή δεδομένων. Αυτό ακριβώς ήταν το ζητούμενο Οπότε τι λέμε εδώ πέρα, ότι η σύγκληση είναι αμοιβαία υποφελής ε, και για την ιδιωτικότητα των ανθρώπων και για την διευκόλυνση του εμπορίου. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα σοβαρό προηγούμενο όταν άλλες μεγάλες χώρες πηγαίνουν σε διαφορετική κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι συμφωνούμε στην σημασία αυτής της ε, απόφασης και θεωρούμε ότι δεν αντικατοπτρίζεται αυτό επαρκώς, κάτι το οποίο ίσως δεν στέλνει το σωστό μήνυμα. Και βεβαίως αυτό το εξτάζουν και οι άλλοι εταίροι μας συγκεκριμένα. Κάποιες επιλεκτικές αναφορές είτε στο Ιαπωνικό δίκαιο είτε στη GDPR ίσως δίνουν την εντύπωση ότι τα δύο συστήματα απέχουν και αυτό αμφισβητεί το επίπεδο προστασίας που διασφαλίζει η Ιαπωνική νομοθεσία. Γνωρίζω πως έχω πολύ λίγο χρόνο. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Παράδειγμα τους κάνει το σχέδιο ψηφίσματα ως ασκή έντονη κριτική το ύψος των προστήμων ε, του Ιαπωνικού συστήματος ε, χωρίς να προβλέπει το ότι προβλέπονται και ποινικέ κυρώσεις μεταξύ των οποίων και φυλάξη. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι ποινικέ ε, κυρώσεις ε, και η φυλάξη είναι οπωσδήποτε παίζουν πολύ πιο αποτρεπτικό ρόλο από τα απλά πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα. Ούτε στην ομολογία του δικαστηρίου, ούτε στο... στην παραπομπή που γίνεται για την επάρκεια των άλλων χωρών δεν γίνεται λόγος για μια αντιστοιχία σημείο προς σημείο, αλλά μιλάει συνολικά για ένα επαρκές επίπεδο προστασίας με άλλα μέσα από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ένωση. Όμως, εάν οι τέτοιες λεπτομερείς συγκρίσεις γίνουν, σας ζητάμε να λάβετε υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλα σημεία που θα μπορούσα να αναφέρω. Ίσως άλλο ένα η ανεξαρτησία της αρχής ε, της Ιαπωνίας, η οποία αμφισβητείται από το ψήφισμα στην παράγραφο 24. Ενώ η ανεξαρτησία αυτή είναι εγγυημένη από την ε, νομοθεσία με παρόμοιες εγγυήσεις που έχουμε και στο GDPR σε σχέση με τους διορισμούς. Τα μέλη της αρχής πρέπει να επιβεβαιωθούν από το Κοινοβούλιο της Ιαπωνίας υπάρχει και προστασία για καταχρηστικές απολύσεις και υπάρχει και η προστασία της ίδιας της ανεξαρτησίας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι χωρίς ε, να υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό επιχείρημα αμφισβητείται αυτή η ανεξαρτησία. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να είμαστε επικοδομητικοί με εταίρους ε, με τους οποίους έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις ε, για να μας ακολουθήσουν και άλλοι σε αυτήν την πορεία. Και νομίζω αυτό είπε και η αντιπροσωπεία της Επιτροπής πέρσι στην Ιαπωνία. Ως συνήθως είμαστε στην διάθεσή σας ε, ακριβώ για να δώσουμε και τις απαραίτητες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, πρέπει να λήξει τώρα η συνεδρίαση κάπου. Προθεσμία για τροπολογίες είναι 21 η Νοεμβρίου. Θα επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αλλάξουμε αίθουσα τώρα. Πάμε στο 3ε2, αν ενδιαφέρεται κανείς ακούσουμε τον κύριο Βάιντεν Χόλτσα. Με τους υπόλοιπους τα λέμε αύριο. Εδώ, ξανά. Γεια σας.